Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Thank you and thank you. Ωραία. Ευχαριστώ και ευχαριστώ εσάς που είσαστε εδώ έγκαιρα. 9 πρέπει να σημαίνει 9, έτσι, γιατί όσοι έρχονται 9, γιατί να κάθονται και να περιμένουν αυτούς που καθυστερούν. Γι' αυτό θα αρχίσουμε. Χαίρομαι που τουλάχιστον κάποιοι είναι εδώ ήδη. Αρχίζουμε με το σημείο 13 στην ημερήσια διάταξη, που είναι ένα σημαντικό σημείο. Πρόκειται για τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης το 2019. Η εισηγήτριά μας είναι η κυρία Στέρντε Λάγκε. Θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης και μετά θα ακούσουμε τους σκιώδες εισηγητές και θα έχουμε και κάτι διά εφόσον έχουμε χρόνο. Ίσως δεν θα πρέπει εγώ να μιλάω εκ μέρους της Εστέρ, εκείνη θα μιλήσει μόνη της. Πάντως αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι δεδομένου του χρονοδιάγραμματος Α, όχι, μετά. Μετά θα μιλήσω εγώ για το χρονοδιάγραμμα και τα λοιπά. Προς το παρόν να ακούσουμε την Έστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, εννέα η ώρα, πίεση, καλά. Αλλά να μπω στην έκθεση. Για σου, από εσά είσαστε νέοι εδώ. Είναι η δεύτερη έκθεση που ετοιμάζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είχαμε για την ετήσια ανάπτυξη και τώρα περνάμε στο δεύτερο που είναι η έκθεσή μας που έχει να κάνει και με τις στάσεις, την υλοποίηση κτλ. Τώρα λοιπόν, συνολικά για την ε, κατάσταση. Θα έχετε ακούσει πολλούς και έχουμε οικονομικές ε, θετικές τάσεις ευτυχώς. Ε, υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία της Ευρώπης ευτυχώς, αλλά υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις ακόμα που έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει ανεργία των νέων σε πολλές χώρες. Ε, βλέπουμε να υπάρχει πίεση στην αγορά εργασίας, να υπάρχουν ε, δυσκολίες σε άλλες χώρες αντίθετα να καλυφθούν κάποιες θέσεις απασχόλησης. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ στην έκθεσή μου είναι ότι υπάρχει και πολιτική αβεβαιότητα. Ας δούμε τον πόλεμο των εμπορικών Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθώ και στους ε, οικονομικούς κινδύνους από το Brexit μετά από αυτά που άκουσα και χτες το βράδυ. Για πολλές χώρες, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, τα στοιχεία δείχνουν ότι θα υπάρχουν προβλήματα. Και μετά, αν δούμε την ε, συνολική εικόνα, μια άλλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η οικονομία μας έχει χαμηλές προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Τώρα δεν θα σας εκπλήξει, όσοι με ξέρετε τουλάχιστον, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναλυφθεί η δράση. σε τρεις πυλώνες, θα έλεγα, που συνδέονται μεταξύ τους. Πρώτα απ' όλα οι δυσημερινομικές πολιτικές, δεύτερον διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τρίτον στρατηγικές επενδυτικές για να ετοιμάσουμε τις οικονομίες μας για τον 21ο αιώνα και τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Αυτό είναι το τρίγωνο που πάντα υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλο πάντων, δεν θέλω να ξοδέψω πολύ από το χρόνο σα, θα αναφερθώ και στα τρία, αλλά κάπω σύντομα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τι δημοσιονομικέ πολιτικές. Εννοείται ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με την όποια ευελιξία έχει ήδη, με πάση περιπτώσει. Πρέπει επίσης να έχουμε οικονομίες αντοχής που να είναι έτοιμες σε περίπτωση νέας ύφεσης και να ετοιμαστούμε επίσης και για το φαινόμενο της γύρανσης του πληθυσμού, το δημογραφικό δηλαδή, το οποίο και αυτό θα πιέσει την οικονομία. Για το θέμα του χρέους, εξακολουθεί το επίπεδο, ο μέσος όρος του επίπεδου χρέου να είναι ιδιαίτερα υψηλό, το οποίο βέβαια διαχειριζόμαστε προ το παρόν μεν, αλλά στο μέλλον μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο. αν η οικονομική κατάσταση, τα επιτόκια αλλάξουν. Τώρα, το fiscal stance. Αυτό ήταν κάτι που μας απασχόλησε πολύ το 2019. Εδώ είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Οι διορθωτικές μεταρρυθμίσεις τώρα. Μπορούμε, πιστεύω, να συμφωνήσουμε όλοι ότι χρειάζονται. Γιατί εφόσον γίνονται με το σωστό τρόπο, βοηθούν τις οικονομίες μας να είναι πιο ανταγωνιστικές και περισσότερο αντοχής. Η αγορά εργασίας επίσης είναι ένα ζήτημα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για μας, προκειμένου στον 21ο αιώνα να μπορέσουμε να έχουμε τα κατάλληλα προσόντα στο εργατικό δυναμικό και βέβαια να γίνονται και κατάλληλες επενδύσεις. Τώρα εδώ βέβαια υπάρχουν διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ των πολιτικών ομάδων όταν ετοιμαζόμασταν για το πρόγραμμα της Επιτροπής, δηλαδή το θέμα της διαβίου, μάθησης, ε, των δεξιοτήτων κλπ. Έρχομαι τώρα στις επενδύσεις. Χρειάζονται για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Χρειάζονται επιπλέον μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το έλλειμμα επενδύσεων που έχουμε διαπιστώσει από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Και εδώ υπάρχουν διαφορές βέβαια ανάμεσα στις χώρες μέλη. Δεν είναι μια λύση που ταιριάζει σε όλους γιατί διαφέρει η κατάσταση από χώρα σε χώρα. Πάντω συνολικά πρέπει να φροντίσουμε ότι θα στηρίξουμε τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, σεβόμενοι βέβαια πάντα τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης. Ε, ξέρετε ότι είναι περιορισμένες οι λέξεις που μπορώ να χρησιμοποιήσω σε μια τέτοια έκθεση, οπότε γι' αυτό έχω περιορίσει και το κείμενό μου. Αλλά αν πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να προσθεθεί, ευχαρίστως θα μπορέσουμε να το προσθέσουμε. Περιμένω τις παρατηρήσεις σας. Τώρα, χρονοδιάγραμμα. Ξέρω ότι είναι σφιχτό. Ε, δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειε αλλά να ξέρετε ότι δίπλα στην πισίνα καθόμουν και έγραφα αυτή την έκθεση. Έγινε, εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμη. Τώρα, γιατί είναι τόσο σφιχτό το χρονοδιάγραμμα. 12 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και αν μπορείτε στα αγγλικά παρακαλώ. Ο λόγος που είναι λοιπόν τόσο σφιχτό το χρονοδιάγραμμα είναι ότι αν θέλουμε το Συμβούλιο να ακούσει τη δικιά μας ε, θέση πρέπει να είμαστε έτοιμοι πριν από την διάσκεψη. Για να μπορέσει η Ολομέλεια δηλαδή να ψηφίσει τον Οκτώβριο, εμείς ε, πρέπει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου στην Επιτροπή μας να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Γι' αυτό και πρέπει να δουλέψουμε το Σεπτέμβριο σκληρά. Εγώ το έκανα. Ε, υπάρχουν κάποιες ε, ώρες που έχουμε προβλέψει για συνάντηση με τους συντονιστές, οπότε ελπίζω με τη δουλειά όλων να τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε. Θα συνοψίσω, Έστερ, στο τέλος το χρονοδιάγραμμα, της προθεσμίες κτλ. Λοιπόν, εκ μέρους των σοσιαλιστών ο Γιώνας θα μιλήσει. Δεν έχουμε το συντονιστή, αλλά θα μιλήσει εκείνο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούκα δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, οπότε εγώ θα διαβάσω αυτό το οποίο ετοίμασε. Εκ μέρους λοιπόν του που ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ σε αυτή την πρώτη συζήτηση, αλλά μεταφέρω όπως σας είπα τις απόψεις της. Πρώτον, θέλει να ευχαριστήσει την εισηγήτρια, την Έστερ για την έκθεσή της. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν ένα υγιές οικονομικό και κοινωνικό κλίμα με πλήρη απασχόληση και με προστασία του περιβάλλοντος. Η Ευρώπη παραμένει η πιο πλούσια ήπειρο στον κόσμο και έχει δυνατότητες για ε, μεγαλύτερη ε, ανάπτυξη συγγνώμη, και επίσης μπορεί να βοηθήσει και στην ενεργειακή μετάβαση. Οι πολίτες πρέπει να έχουν θέσεις απασχόλησης η οικονομία αλλάζει γρήγορα και πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές, ώστε οι εργαζόμενοι να μην είναι, όπως γίνεται συνήθως, τα πρώτα θύματα. Η ομάδα μας, λοιπόν, προτείνει διάφορες τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την αύξηση των επενδύσεων, κυρίως όσον αφορά την οικολογική μετάβαση, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και σταθερότητα των τραπεζών και καταπολέμηση των ανισοτήτων με κοινωνική δικαιοσύνη. Ελπίζω, λέει, η συγγήτρια να μπορέσει να συμπεριλάβει τις ε, τροπολογίες μας ε, στο κείμενο. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Περνάμε στον επόμενο. Όλιβερ Σεστέλ από το Ρινιού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο σκιώδης μας δεν είναι εδώ. είναι μια έκθεση πάνω στην οποία προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία με την κυρία Λάγκε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα άλλο. Εμείς είμαστε νέα ομάδα, ε, νέοι ευρωβουλευτές. Συγγνώμη γι' αυτό. Okay, so... Καλώς. Πράσινη, δεν έχουμε εισηγητή, αλλά Σβέν. Ε? Ναι. Ε, ευχαριστώ εκ μέρους. Ε, του εισηγητή μας που ορίστηκε αυτή την εβδομάδα μόνο. Ο κύριος Ορτασούν είναι. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι εκ μέρους του να αναφέρω κάποιες παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε για το σχέδιο έκθεση στην εισηγήτρια. Έχουμε δει τις ε, συστάσεις Επιτροπής και έχοντα και μακρά εμπειρία από τέτοιου είδου εκθέσεις, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βεβαίω στην έκθεσή σας υπάρχουν πολλά σημαντικά με τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε, όπως για παράδειγμα το πόσο λίγο οι χώρες ακολουθούν τις συστάσεις. Η αξιολόγηση, μάλιστα εγώ θα έλεγα, παρένε θετική, γιατί τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, θεωρούν ότι υπάρχει κάποια πρόοδος. Αν δει κανείς τη συνολική πρόοδο θα καταλάβει ότι οι χώρες μέλη ελάχιστα υλοποιούν, ελάχιστα παίρνουν στα σοβαρά. Τελικά είναι οι χώρες οι οποίες αποφασίζουν για τις συστάσεις. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ανοιχτό και να μην ακολουθήσει την αξιολόγηση και τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι είναι πρόοδος. Γιατί εμεί δεν θεωρούμε ότι υπάρχει αρκετή πρόοδος. Έπειτα, διαφωνούμε και γενικά για το οικονομικό μείγμα πολιτικής. Εμείς κυρίως επειδή σε μία από τις πιο μεγάλες περιόδους οικονομικής ανάπτυξης έχουμε μείωση της ανεργίας και των ελλημάτων, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά το να λέμε ότι είναι επειδή έχουμε υιοθετήσει πάρα πολύ καλές ε, πολιτικές δεν είναι πολύ αξιόπιστο δεν είναι επειδή οι χώρες μέλη κατάφεραν να συνεργαστούν τόσο καλά για να δημιουργήσουν την έννοια αγορά, αλλά επειδή συνολικά υπήρχε μακροοικονομικά σταθερότητα. Άρα και εδώ πρέπει να είμαστε επικριτικοί. Πρέπει να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη δράση από τη δικιά μας την πλευρά για να έχουμε μια καινοτόμο, σταθερή και αναπτυσσόμενη ενιαία αγορά. Έπειτα το θέμα του περιβάλλοντος έχει ξεφύγει το καλοκαίρι από το μυαλό της εισηγήτριας από ό,τι φαίνεται. Θα έπρεπε όμως να περιλαμβάνεται σε μια τέτοια έκθεση. Και δεν θα έπρεπε να πρόκειται για τροπολογία, θα έπρεπε να βρίσκεται στον κορμό του κειμένου Οπότε, ναι, λέτε υπάρχει δυνατότητα για ανάπτυξη, ναι, αλλά και για πρασίνισμα. Και σε μια τέτοια έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται αυτό, να είναι ορατό. Τέλος, έχουμε και κάποια προβλήματα με τις διάφορες ανισορροπίες. Ο όρος φτώχεια δεν υπάρχει στο σχέδιο. Υπάρχει όμως την αρχική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή επίσης στις συστάσεις προς διάφορες χώρες έχει αναφέρει τον επιθετικό ανταγωνισμό και για τις κάτω χώρες. α, ναι, σωστά. Και Μάλτα, ναι. Και Μάλτα, εδώ είναι στην αίθουσα. Λοιπόν, πολλές χώρες για πρώτη φορά ή για δεύτερη φορά στις αναχώρα συστάσεις ε, είχαν τέτοια σχόλια. Αυτό λοιπόν πρέπει να σημειωθεί και να επικρίνουμε τις χώρες μέλη που έχουν κάνει ελάχιστες ε, προσπάθειες για να αποφεύγουν τον επιθετικό ανταγωνισμό. Και νομίζω ότι είναι κάτι με το οποίο πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε, ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό χώρο προερχόμαστε. Ελπίζω λοιπόν να τα καταφέρουμε και να μην γίνει ένα νέο επεισόδιο μακροοικονομικών συγκρούσεων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η έκθεση, αλλά αντίθετα να γίνει μια έκθεση αποδεκτή από το ευρύ φάσμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γκούναρ Πεκ δεν είναι εδώ. Άλλος κανείς. Ποιος, εσείς. Δεν έχουμε κανέναν από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ωραία. Από το ECR έχουμε εδώ κάποιον. Εσείς, εκ μέρους του ECR. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Σλοβακικά θα μιλήσω. Συνεπώς, κυρία εισηγήτρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υποβάλλατε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Πιστεύω ότι η εισηγήτρια έχει κάνει καλή δουλειά. Κύριε Λάγκε, συμφωνώ με το πνεύμα της έκθεσής σας. Κυρίως που λέτε ότι σε καλούς καιρούς πρέπει να αποταμιεύουμε, να ε, προστατεύουμε, να παγιώνουμε ε, τα οικονομικά μας σε καλούς καιρούς πρέπει να το κάνουμε αυτό πράγματι, γιατί μετά τους καλούς καιρούς έρχονται κακοί καιροί και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ένα πράγμα θα πρόσθετα, το δημόσιο χρέος. Είναι καλύτερα να γίνεται εξυγίανση παρά να μιλάμε για μεγάλα ταμεία. Όταν μιλάμε δηλαδή για την προετοιμασία για χειρότερες εποχές. Επίσης, στο σημείο 8 που μιλάτε για μεταρρυθμίσεις, εδώ ανταγωνισμός που θα βοηθήσει να εξηγενθούν τα δημοσιονομικά. Επίσης, σύμφωνα και για τα θέματα για τις μεταρρυθμίσεις. Τώρα, στα σημεία 12 με 14 που αναφέρονται στις επενδύσεις. Εδώ λέμε ότι η Ευρωζώνη έχει πολύ χαμηλές επενδύσεις. Χρειάζεται να έχουμε περισσότερες επενδύσεις στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Εδώ δυστυχώς πρέπει να πω ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι σημαίνει πολλές επενδύσεις και τι σημαίνει λίγες επενδύσεις. Η πρόταση αυτή φαίνεται ελκυστική, αλλά μην ξεχνάμε ότι το επίπεδο πριν από την κρίση ήταν ένα θέμα το οποίο οδήγησε στην κρίση. Οπότε, όταν είμαστε σε ανάπτυξη να επενδύουμε, δεν ξέρω, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι ε, απόδοση έχουν αυτές οι επενδύσεις και πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις πάντα για μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Μέσα σε αυτό το πνεύμα θα υποβάλουμε και εμείς τις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γκουέ. Χωσέ Γκουσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα μιλήσω πορτογαλικά. Πιστεύω ότι η συζήτηση που κάνουμε εδώ για την έκθεση αυτή, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί για τις διαφορές μεταξύ μας, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα που αναφέρονται στην έκθεση και που είναι το τζάργον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής πρώτα απ' όλα. Μια τέτοια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να αναφέρεται και στην οικονομική βιωσιμότητα, εννοείται, αλλά και για μας δεν είναι αντιφατικό αυτό, θα πρέπει συγχρόνως να ανταποκρίνεται στους μεγάλους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή μετάβαση είναι όροι που έχουν μπει στις εκστρατείες όλων των κομμάτων, όλων των χωρών και είναι και οι αποφάσεις που παίρνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζουμε σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν τελικά αντίκτυπο στη δημοσιονομική μας πολιτική. Οπότε το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τη φτώχεια και για την ε, απασχόληση. Δεν είναι αντιφατικά όλα αυτά. Η έκθεση αναφέρεται στην εξέλιξη των δικτών όσον αφορά το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη δικιά μου τη χώρα για αυτά τα θέματα υπήρξε μεγάλη μείωση και βασίζεται στην μείωση των ε, μισθών. Οπότε πρέπει να δούμε πώς εξισορροπούνται όλες αυτές οι πολιτικές. Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσουμε και το θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Είναι και αυτός ένας όρος ε, της ευρωπαϊκής τζάργων, αλλά τι ακριβώς σημαίνει. Πολλές φορές ο όρος αυτός χρησιμεύει για να δημιουργείται συνένεση, συμφωνία μεταξύ πολιτικών δυνάμεων που στην ουσία έχουν διαφορετικές απόψεις για την αγορά εργασίας. Τελικά όμως εμποδίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρει ουσιαστικά στη συζήτηση. Γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι το Συμβούλιο ακούει για διορθωτικές ε, μεταρρυθμίσεις από την Επιτροπή και τελείωσε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Να δούμε ε, το θέμα της αγοράς εργασίας, για παράδειγμα. Και θα έπρεπε να αναφέρεται αυτό με κάποιο τρόπο στην έκθεση. Έπειτα τις ε, αναχώρα συστάσεις. Δεν είναι τόσο ειδικέ αναχώρα. Εξαρτάται φυσικά για ποια χώρα μιλάμε. Πάντως, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε ότι είναι ικανοποιητική η κατάσταση, δεν ξέρω γιατί υπάρχουν πληροφορίες αντιφατικές. Αλλά αν δεν είναι ικανοποιημένοι από την εφαρμογή των συστάσεων, το πρόβλημα ίσως δεν είναι το πρόβλημα της χώρας, αλλά το πρόβλημα των συστάσεων. Οι συστάσεις ίσως δεν ανταποκρίνονται καλά στην κατάσταση. Γιατί αν έχουμε μία αδύναμη περιοχή, αυτό οφείλεται στην νομισματική πολιτική. Δεν έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε εδώ. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια και εμείς Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε επικοδομητικά μαζί της. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Είναι σημαντικό να έχουμε τώρα και το Catch Όχι μόνο γιατί έχουμε χρόνο, αλλά γιατί είναι και ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Θα βασιστώ στη σειρά με την οποία ζητάτε το λόγο. Η Μαργαρίτα Μάρκες πρώτα από τους σοσιαλιστές. Και μετά η κυρία Φιγκέιρα από το Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και θέλω να σας πω ότι έχω να κάνω κάποια σχόλια για την έκθεσή σας. Το πρώτο αφορά την έννοια, τον όρο, τους ορισμούς τις ε, χώρες οι οποίες είχαν ε, τρόικα στις χώρες οι οποίες είχαν τρόικα, οι μεταρρυθμίσεις, οι διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, τέθησαν σε κίνδυνο. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα της επενδύσεις, εκεί υπάρχουν ε, δύο θέματα που πρέπει να βάλουμε σε αυτό το θέμα των επενδύσεων. Το πρώτο είναι επενδύσεις για να υπάρχει σύγκληση και επίσης χρειαζόμαστε και επενδύσεις για τη μετάβαση σε οικονομία χωρίς άνθρακα και σε ψηφιοποιημένη οικονομία. Πολλές φορές το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, εγώ παλαιότερα ήμουνα μέλος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, εκεί συζητήσαμε πάρα πολύ σχετικά με το ότι τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να οικειοποιηθούν περισσότερο το CSR. Τα κράτη-μέλη, στη τελική ανάλυση, αντιδρούν και οι συστάσεις είναι συστάσεις ε, που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. το πώς τα κράτη-μέλη δέχονται τις συστάσεις, αυτό δεν αρκεί. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πείσει τα κράτη μέλη να οικειοποιηθούν περισσότερο, να θεωρήσουν διοκτησία τους το θέμα ε, των συστάσεων. Καλημέρα σας. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ ε, που είναι σε μακροοικονομικό επίπεδο, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα που νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι το Brexit. Βεβαίως όλες οι χώρες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις επιπτώσεις από το Brexit, είτε υπάρχει ε, συμφωνία, είτε γίνει αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Και αυτό θα πρέπει να ενταχθεί ως στοιχείο στους ε, προϋπολογισμούς μας και στον οικονομικό προγραμματισμό. Το δεύτερο που θέλω να πω ε, σε σχέση με την στέγαση. Βλέπουμε ότι μία κρίση στέγαση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, οικονομία μας και για μας τους πολιτικούς ε, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, κρίσης αυτής. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε όλο και περισσότερο ε, τα διάφορα εργαλεία που υπάρχουν σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και νομίζω ότι τελικά αν το θέμα δεν το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά θα προκύψει κρίση. Το τρίτο που θέλω να πω έχει σχέση με τους στόχους της χιλιετίας. Εχθές ε, στην Επιτροπή ΝΤΕΒΕ ακούσαμε μία θαυμάσια εκθέση σχετικά ε, με τις ε, επενδύσεις που χρειαζόμαστε εάν αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους της χιλίτιας. Νομίζω ότι μπορεί κανείς το θέμα να το δει και κάτω από διαφορετικό πρίσμα όμως εκείνο που παίζει ρόλο είναι η ποιότητα ζωής, αλλά εκείνο που παίζει επίσης ρόλο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου τους στόχους της χιλιετίας, ε, ειδικά ιδιωτικέ επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ χαμηλές, γύρω στο 16%. Πρέπει αυτό να το εξετάσουμε. Και τέλος, όσον αφορά στην ανάπτυξη, πραγματικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το στοιχείο του φίλους και των προοπτικών. Γιατί αν δούμε λιγάκι ε, το θέμα της ψηφιακής αγοράς, θα διαπιστώσουμε ότι ο αποκλεισμό των γυναικών είναι τεράστιο οικονομικό θέμα, ε, διότι στις οικονομίες μας συμμετέχουν όλο και λιγότερες γυναίκες σε θέματα που αφορούν στην ε, πληροφορική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πολύ σημαντική δουλειά της και όπως ε, το έκαναν και οι προλαλήσαντες και εγώ ε, θέλω να αναφερθώ στο πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά τα οποία εξετάζουμε. Και ξεκινάω από την παραδοχή που αναφέρεται σε αυτή την έκθεση ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. Υπάρχουν ε, οι βασικές αρχές ε, που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια τέτοια βασική αρχή είναι και η αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αν δώσουμε σημασία μόνο στην ανταγωνιστικότητα, αυτή δεν είναι μια σωστή μέθοδος ε, κατά την άποψή μου γιατί ε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το ότι θα υπάρχει σε όλα τα κράτη η ίδια ανάπτυξη και ομοιογενής ανάπτυξη. Έχουμε διαπιστώσει παλιμένα ότι αυτό το θέμα της ανταγωνιστικότητας έχει προκαλέσει ανηλεή ανταγωνισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη και σε τελική ανάλυση που καταλήγουμε. Καταλήγουμε ότι ένα κράτος ενδεχομένως να παρουσιάζει μια τεράστια ανάπτυξη, αυτό όμω εις βάρος της ανάπτυξης άλλων κρατών. Και αυτό το διαπιστώσαμε κυρίως ε, όσον αφορά τις, ε, τη διαφορά που υφίσταται ανάμεσα στις ε, χώρες του Βορρά και στις χώρες του Νότου, γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία εγώ συμμερίζομαι απολύτως και υπάρχει και το θέμα των ε, ε, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και εκεί υπάρχουν ε, οι ίδιοι προβληματισμοί, γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι η ποιότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων, η ποιότητα αυτή μεταβιβάζεται πλήρως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδαμε τι έγινε με την Ελλάδα. Έχουμε εμπειρία από την Ελλάδα. Οι μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε κοινωνική καταστροφή, σε καταστροφή στο θέμα της απασχόλησης, στη ζωή, ε, στη κοινωνικά εχέγγυα που χρειάζονται οι πολίτες, άρα δηλαδή μεγάλη κρίση της δημοκρατίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ψήφος ε, των πολιτών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταδείξει ότι αντιτίθενται πολίτες ε, σε τέτοιου είδους ε, πολιτικές. Όμως δεν άλλαξε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα και τότε που ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ, αναγνώρισε το γεγονός ότι αυτές οι πολιτικές λιτότητας και αυτές οι πολιτικές μεταρρύθμισης, κυρίως όταν πρόκειται για αυστηρές πολιτικές μεταρρύθμισης, ε, αυτές οι πολιτικές δεν βοήθησαν τελικά στην ανόρθωση της οικονομίας τουλάχιστον της Ελλάδας. Το να επιμένουμε λοιπόν σε αυτή την γραμμή, σε αυτή την πολιτική την οποία αμφισβητούν ε, οι περισσότεροι οικονομολόγοι, μια πολιτική που κατά την άποψή μου οδήγησε στο να αναχαιτιστεί η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, ε, αυτό δεν είναι σωστό. Εγώ πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι κυρίως ανάμεσα, αν θέλετε, στην Ευρωζώνη και άλλες ε, χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Είναι δύσκολο, όπως σας είπα, να υπάρξει ομοιογενής και σταθερή ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της ε, Ευρωζώνης. Και μόνο αυτό, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου και τις παγκόσμιες προκλήσεις, τα σόκα τα οποία αντιμετωπίζουν τα συστήματά μας. Με λίγα λόγια θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οφείλουμε να έχουμε κατά νου την αρχή της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων θέματα τα οποία είναι παγιωμένα στις, στα συντάγματα των κρατομελών και δεν μπορούν να παραγνωρίζονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλος ένας ομιλητής από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είπε ο πρόεδρος από την Ελλάδα, για Ε, εχθές ε, ακούσαμε ότι η νομισματική πολιτική θα συνεχιστεί και αυτή θα επηρεάσει την ανάπτυξη διότι ε, χρηματοδοτείται από τα αρνητικά επιτόκια των ε, ε, πολιτών. Υπάρχουν λοιπόν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις η αναχρηματοδότηση του χρέους τελικά είναι χαμηλότερη και επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτή την ανώμαλη νομισματική πολιτική. Οι ε, δημοσιονομικές ισορροπίες επίσης επηρεάζονται. Εγώ Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την ε, νομισματική πολιτική στην οποία βρισκόμαστε. Ε, θα ήθελα να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και θέλω να ελπίζω ότι τη συζήτηση αυτή θα την έχουμε και με την κυρία Λαγκάρτ αλλά και με άλλους ε, θεσμούς όταν θα συζητήσουμε το οικονομικό και νομισματικό μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν βλέπω να υπάρχει άλλος στη διαδικασία Catch the Eye. Ε, να κάνω δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι ε, εγώ δεν συμμερίζουμε απαραίτητα την υπερβολική απεσιοδοξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βεβαίως και έχουμε χάσει χρόνο, ε, κυρίως ε, τότε που ήταν εύκολο να γίνουν ταχείες αλλαγές και σε χαλεπούς καιρούς τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Γνωρίζουμε καλά ότι πολλά βρίσκονται στα δικά μας τα χέρια και Παράλληλα όμως γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κάνει και η έκθεση. Εκτιμώ αυτά που είπε ο Σβέν. Ε, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει σε θέματα που είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την πίεση, ε, πρέπει να ασκήσουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη πίεση. Αυτός είναι ο στόχος της έκθεσης. Ε, παρακαλώ, Εστέρ, εσείς μπορείτε να ανακεφαλαιώσετε. Yes, thank Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, Πρόεδρε, και μετά από αυτά που μας είπατε και προηγουμένως, ε, αυτό αναφέρθηκε και σε διάφορες ε, παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τις συστάσεις χώρα. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα θα πρέπει να βρούμε μία διατύπωση. Και καταλαβαίνω ότι οι σοσιαλιστές στέλνουν διαφορετικά κάπως μηνύματα, να το θέσω έτσι. Μ' αρέσει το σχόλιο του Σφέντσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως να τα βλέπει όλα πολύ ρόδινα και ενδεχομένως ότι η μερική συμμόρφωση με τις συστάσεις σε ένα χώρα δεν σημαίνει πλήρη συμμόρφωση, καταλαβαίνω τι λέει, σε ό,τι αφορά το θέμα ιδιοκτησία. Αυτό, ναι, συχνά το ακούμε στην συζήτηση. Από την άλλη, δίνεται μέγιστη ευελιξία στα κράτη-μέλη προκειμένου να δράσουν με τον τρόπο που θεωρούν τον πλέον ενδεδειγμένο. Και άρα για να βγαίνουμε και να λέμε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διεκτησία, όχι. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συμμόρφωση. Όταν θέτουμε το θέμα τη ιδιοκτησία. εντάξει, είναι διαφορετικό το γεγονός όμως ότι μόνο, ότι μόνο οι σύμβουλοι δίνουν την αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη να δράσουν όπως πρέπει, έτσι θα δημιουργηθεί η ιδιοκτησία. Άρα εδώ πέρα θεωρώ ότι τίφεται θέμα ερμηνείας και υπάρχουν κάποιες διαφορές με τους πράσινους, αλλά μπορούμε, θεωρώ, να βρούμε κάποιο κοινό σημείο ξεκινάμε όμως με αυτό που είπε ο Σβέν. Δεν είναι η μερική συμμόρφωση, πλήρη συμμόρφωση. Σε ό,τι αφορά τώρα το δυναμικό απασχόληση, σε ό,τι αφορά τη μεταβάση της ενέργειας, ε, τις ε, επενδύσεις στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα. Αν επικεντρωθούμε στο δυναμικό απασχόληση όπω το διατυπώσατε, είναι ενδιαφέρον θεωρώ. Ε, τίθεται το θέμα της ανταγωνιστικότητας στη συνέχεια, το είπα και εισαγωγικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο έχει χαμηλό δυναμικό ανάπτυξη σε σχέση με τους υπόλοιπους και αυτό που θεωρώ ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Αν ο γιος μου, ο οποίος είναι 16 τώρα, ε, πρέπει να βγει στην παγκόσμια αγορά και να συναγωνιστεί με τους υπόλοιπους, θα ήθελα να συναγωνιστεί όχι μόνο βάσει τιμής. Δεν πρόκειται ποτέ να είμαστε πιο φθηνοί. Πάντα θα υπάρχουν φθηνότερα χέρια από τα ευρωπαϊκά. Άρα, αν δεν θέλω λοιπόν αυτό να είναι το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, θα πρέπει η Ευρώπη να είναι πιο έξυπνη, η πρώτη σε πολλού τομεί. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε καινοτομία. Και η καινοτομία συχνά προωθείται από την ανταγωνιστικότητα. Δεν μιλάω για μια ανταγωνιστικότητα μέχρι τελικής πτώσης μεταξύ των κρατών μελών, αλλά με ανησυχεί το συνολικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα μεγάλο θέμα, μια μεγάλη πληγή και θεωρώ ότι το θέσατε εύστοχα. Φράνσις, για το Brexit. Μου άρεσε η διατύπωσή σας ότι θα πρέπει να το βάλουν τα κρατημέλη στο μελλοντικό προγραμματισμό τους. Ακόμα και αν είναι από την ομάδα μου, φυσικά να κάνετε τροπολογίες για τη στέγαση. το θέμα επικουρικότητας, προφανώς, αλλά αν συμμετέχετε σε άλλο επίπεδο άσκησης πολιτικής πέρα από το ευρωπαϊκό, ξέρετε ότι το θέμα αυτό είναι μεγάλο. Έχει ευρωπαϊκούς και εθνικούς ευρωπαϊκέ και εθνικέ συνιστώσει στο θέμα αυτό. Και ενδεχομένω κάποιε κυβερνήσει να θέλουν να το αντιμετωπίσουν ω τέτοιο. Το θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη, του ΣΒΕΝ, σχετίζεται με την ε, δυνατότητα απασχόληση, το δυναμικό απασχόληση σε, σε πολλού τομεί. Νομίζω ότι α, αναφέρθηκα στα πιο πολλά θέματα. Το τελευταίο θέμα σε ό,τι αφορά την νομισματική διάσταση θεωρώ ότι είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο ακούγεται πολύ και στην δική μου χώρα. Αν το κάνουμε copy-paste στην έκθεση αυτή δεν θα είμαστε έτοιμοι πριν το Οκτώβριο, πριν τη σύνδεση τον Οκτώβριο. Αλλά αναφέρω το κόστος του χρέους, το οποίο σχετίζεται με τη συζήτηση που θίξατε και μια προειδοποίηση επίσης ότι θα αυξηθεί το κόστος για την εξυπηρέτηση του χρέους στο μέλλον. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο μπορούμε να αναπτύξουμε το σκέλος αυτό. Νομίζω ότι αναφέρθηκα στα πιο πολλά στοιχεία. Και προσβλέπω στην πρώτη συνεδρίαση των συντονιστών στο Στρασβούργο, αν δεν κάνω λάθος, καλά τα λέω γραμματεία. Στο Στρασβούργο δεν είναι η πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών. Ναι, ναι, ναι, λέει ο πρόεδρος. Να συνοψίσω. Γιατί υπάρχουν κάποιες συνέπειες της μετάθεσης του θέματος στην Σύνοδο του Οκτωβρίου. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα ATM για την, τις τροπολογίες και άρα σας ζητούμε να καταθέσετε τις τροπολογίες γραπτά σε έγγραφο Word, δηλαδή στα αγγλικά, αν γίνεται, για να μπορέσουμε να κάνουμε τους συμβιβασμούς. Αν χρειάζεστε, θα σας βοηθήσει η γραμματεία. Προθεσμία για τα κατάσταση τροπολογιών. 12 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Και να έχετε υπόψη σας ότι δεν χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό σύστημα, επαναλαμβάνω. Επίσης, συνάντηση με τα Αθηνικά Κοινοβούλια 24 το απόγευμα, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 2 ή 3 Οκτωβρίου και ελπίζουμε στην 1η του Οκτωβρίου να ψηφιστεί το θέμα στην Ολομέλεια. Σκιώδης 18 στο Στρασβούργο και άλλες ε, τρεις συναντήσεις μεταξύ της, μετά τις 23 του μηνός. Να σας υπενθυμίσω ότι είναι σημαντικό να περάσει από την Ολομέλεια όπως έχει προγραμματιστεί το θέμα. Αυτό σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Να κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών και τα λέμε στις 10 για το επόμενο θέμα. interesting. So, dear colleagues, please get seated. We, we start. Καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι. So we have now point number... Είμαστε λοιπόν τώρα πλέον στο σημείο 14, ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σχετικά με την κατάσταση εφαρμογή τη νομοθεσία για την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων. Ένα αντιδικαστικό πρόεδρο, επιτρέψτε μου. Να παρατηρήσω ότι όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι ο Πρόεδρο τη Επιτροπή μα διορίστηκε Υπουργό Οικονομικών στην Ιταλία και θα ήθελα να προτείνω να στείλουμε τα συγχαρητήριά μας ως Επιτροπή. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, βεβαίως μπορούμε να αποστείλουμε τα συγχαρητήριά μας ως Επιτροπή. Και να σας πω ότι προγραμματίζουμε την Δευτέρα το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, μετά τη συνεδρίαση του Στρασβούργου, να γίνει στη συνεδρίαση μάλλον της ομάδος το θέμα αυτό να Να περάσουμε λοιπόν στην αλλαγή απόψεων. Να συζητήσουμε την ε, οδηγία και τις περιπτώσεις νομιμοποίησης εισόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Το έχουμε συζητήσει και στην προηγούμενη θητεία, μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και την Danske Bank και τις ε, επαφέ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Απρίλιο του 2019 η ε, Ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών ξεκίνησε έρευνες για την Δανία και την Ρετονία ε, σε ό,τι αφορά ε, τις εστονικές τράπεζες και το Danske Bank. Και η το Συμβούλιο της ΕΜΠΑ απέρριψε τι θέσει και τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση του Κοινοβουλίου για την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση της, του ξεπλήματος χρήματο. και αυτό συνοδεύεται από τέσσερι εκθέσεις για την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο από εγκληματικέ ενέργειες που επιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση. Ε, έχετε στη σελίδα αυτή τα σχετικά στοιχεία. Κατά δεύτερον, το πλαίσιο για την ε, χρηματοοικονομική ευφυΐα, για ε, καλύτερη συνεργασία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, εκτίμηση των συνθήκων για την πιο ασφαλή την πιο ασφαλή μητρώα. Τέταρτο σύστημα τέτοια έκθεση σε ό,τι αφορά το σύστημα της κατηγορίας για καταχρήσεις από ευρωπαϊκές ε, υπηρεσίες. Πρόκειται λοιπόν για την πρώτη παρουσίαση του κυρίου Δεκάμπα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Η Επίτροπος Γιούρεβα προσκληθήκε, αλλά δεν μπορούσε να παραβρεθεί για προσωπικούς ε, λόγους. Την εκπροσωπεύει η Αλεξάνδρα Γιούρ Χρέντερ η οποία είναι υποδευθυντής της DG Just. Θα έχουμε 5 έως 7 λεπτά για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Μετά θα ακολουθήσουν 5 έως 7 λεπτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά θα έχουμε ένα γύρο απαντήσεων και αν υπάρξει χρόνος θα υπάρξει και διαδικασία Catch the Eye και θα σας ζητήσω συγγνώμη που θα φύγω τη μέση της κουβέντας της συζήτησης γιατί έχω αντλημένες υποχρεώσεις και θα καλέσω τον ε, συναδέλφο. Και να δώσω λοιπόν το λόγο στον συναδέλφο, στον ε, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Αρχής Τραπεζών. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετέχω στη συζήτηση. Αξιότιμοι βουλευτές, θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε τρεις αρχές. Τι κάναμε στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εισόδων από κλιματικές δραστηριότητες. Κατά δεύτερον, η βραχυπρόθεσμη προοπτική που έχουμε για τη δουλειά μας σε ό,τι αφορά και την, ε, τις νέες ε, αρμοδιότητες που έχουμε και κατά τρίτον μια ευρύτερη αξιολόγηση του τομέα της καταπολέμησης νομιμοποίησης εισόδων από κλιματικές δραστηριότητες και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στο μέλλον. Όπως ξέρετε, μαζί με τις υπόλοιπες σε αρμοδιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα στο ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα, χρηματοοικονομικό σύστημα και έχουμε νομική ε, υποχρέωση να εφαρμόσουμε σωστά την ε, σχετική οδηγία. Αυτή η εντολή τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιηθεί σε τρεις τομείς ε, στην πολιτική, αναθεώρηση της υλοποίησης από τα κράτη-μέλη και στον τομέα της ερευνά ε, συγκεκριμένων περιπτώσεων σε ό,τι αφορά τη σωστή εφαρμογή της ε, νομοθεσίας. Και έτσι έχουμε συλλέξει εμπειρίες ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε μοιραστεί αυτές τις εμπειρίες μας αυτές και γι' αυτό καλώς ορίζουμε την τελική έκθεση την οποία ανέφερε ο Πρόεδρος, όπου εντοπίζονται κάποια στοιχεία και η οποία δημοσιεύτηκε πέρυσι τον Ιούλιο. Για να σας πω κάποια από τα πορίσματα της έκθεσης. προκλήσει σε ό,τι αφορά τα αποτελεσματικά συστήματα, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαφορέ μεταξύ των συστημάτων διαχείριση κινδύνου σε ό,τι αφορά τον τομέα αυτό. Πιο σημαντικό επίση, μια και είμαστε εποπτική αρχή, μαζί με τι υπόλοιπε εποπτικέ αρχέ, παρατηρούμε ότι υπάρχουν σιγά σιγά καλές πρακτικές, οι οποίες ε, έχουν να κάνουν σε ό,τι αφορά την προσέγγιση κινδύνου για τα ζητήματα αυτά και έχουν να κάνουν σε κάποιες περιπτώσεις με την ε, σωστή ή μη εντολή. Υπάρχουν επίσης πολύ διαφορετικές εθνικές προ, ε, προσεγγίσεις ε, των υποπτικών αυτομέτρων και ότι απιστώνουμε ότι συχνά είναι πολύ προορισμενη η συνεργασία μεταξύ των αρχών, ιδιαίτερα στις συνοριακές ε, δράσεις. Ε, διασυνοριακές δράσεις. Ε. Για τις προκλήσεις. Έχουν γίνει κάποια λάθη στο παρελθόν και νομίζω ότι αξίζει να τονίσουμε ότι τα βήματα που έχουν ληφθεί για την διόρθωση των συστημάτων αυτών έχουν αποφέρει καρπούς. Υποστηρίζουμε λοιπόν την προσέγγιση βάση κινδύνου σε ό,τι αφορά τη χρηματοδοτήση, τους ελέγχους και την εποπτεία. Ενθαρρύνουμε καλύτερο συντονισμό να διευκρινιστούν οι διαφορετικοί ρόλοι σε ό,τι αφορά την εποπτεία και σε ό,τι αφορά τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Συνεργαστήκαμε και με τις υπόλοιπες ESA, τις εποπτικές αρχές, για να αναπτύξουμε κατευθυντήριες γνώμες για τους ποιοι θα είναι οι παράγοντε που θα επηρεάσουν την διαχείριση κινδύνου, για την εποπτεία των ε, ε, περιπτώσεων νομιμοποίησης εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και νομίζω ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ό,τι έχουμε κάνει είναι κατευθυντήριες γραμμές. Αυτά είναι τα εργαλεία που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας, ε, δεδομένου και του πλαισίου της νομοθεσίας στην οποία λειτουργούμε. Δεν είναι φυσικά δεσμευτικά και άρα δεν είναι και πολύ... Είναι μάλλον αδύναμα εργαλεία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση τώρα κάνουμε εκπαιδεύσεις, καταρτήσεις ε, για να προωθήσουμε τη συνεργασία. Έχουμε ένα πολιτές πρόγραμμα εφαρμογής ε, όπου αξιολογούμε τις, ε, την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας από τις εθνικές αρχές. Σας είπα ότι έχουμε στην εργαλειοθήκη μας την δυνατότητα στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος, να κοιτάξουμε την περίπτωση της Μάλτας. Επίσης αναφέραμε και κάτι εισαγωγικά στην περίπτωση της Εστονίας και της ε, Δανίας. Δεν διαπιστώσαμε παραβίαση του κοινωτικού δικαίου στις περιπτώσεις αυτές. Να πω ότι γίνεται επίσης έρευνα για θέματα επίσης ε, AML σε ό,τι αφορά έρευνε οι οποίε θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλο του ε, έτου. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο μέλλον, τι έχουμε στην ατζέντα μα. Και αυτό αποτελεί αποτέλεσμα τη σχετική ε, έκθεση. Ε, Καταρχά, έχουμε αποκλειστική ερμοδιότητα στο θέμα αυτό. Όχι κοινή ερμοδιότητα με τι άλλε εποπτικέ αρχέ, είναι να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή τη οδηγία AML στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπω σα είπα, θα πρέπει να συντονίσουμε ε, την ε, παρακολούθηση της υλοποίησης. Έχουμε λοιπόν τρία άτομα τα οποία εργάζονται με πλήρη απασχόληση στο θέμα αυτό και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και άλλα μέλη που θα προσθεθούν στην ομάδα μας. Είναι ενθαρρυντικό αυτό. Να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε άλλα πέντε άτομα τουλάχιστον για το επόμενο έτος. Έχουμε πολύ περιορισμένους ε, πόρους. Τι θα κάνουμε στο μέλλον. Θα αναπτύξουμε τη συνεργασία και να παρακολουθούμε την ε, υλοποίηση σε σκέλος του συντονισμού θα κοιτάξουμε τις ε, κατευθυντήριες γραμμές θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν αποπτικά συμβούλια ML ε στο εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι το αντίστοιχο που υπάρχει και στην τραπεζική εποπτεία. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια σώματα εποπτεία τα οποία είναι ε, τυποποιημένα στη φύση του, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση αυτή και επίσης ε, κάποιες ε, τράπεζες ε, πολυεθνικές θα έχουν τέτοια αρμοδιότητα να παρακολουθούν τακτικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση τη οδηγία AML και να υποβάλουν εκθέσεις για το ποιο, πώς έχει κατάσταση και πώς εξελίσσεται. Θα συνεχίσουμε και θα βελτιώσουμε την παρακολούθηση και τις εκτέσεις εφαρμογής από τις αρχές. Θα περιλαμβάνετε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας από πλευρά των αρχών για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με θα κάνουμε διμερείς ε, συζητήσεις με τις αρχές και για να βρούμε πού είναι οι αδυναμίες και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και επίσης ε, σκοπεύουμε να κάνουμε και αξιολογήσεις ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εντοπίσουμε τα κοινά σημεία αδυναμίες που χρειάζονται κοινή δράση. Τέλος, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα υποβάλλουμε κατευθυντήριε γραμμέ για να ενισχύσουμε του μηχανισμού εποπτεία των διαφόρων αρχών. Ελπίζουμε να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση με τι ε, οδηγίε αυτέ. Γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά. Ε, ένα λεπτό μου μένει να σας πω τι θα κάνουμε στο μέλλον και ποιε θα είναι οι βασικές μας προκλήσει. Πρόσφατα έχουν γίνει σημαντικέ αλλαγέ σε ό,τι αφορά την οτροπία που επικρατεί για τι δραστηριότητε χαμηλού κινδύνου σε ό,τι αφορά δραστηριότητε AML. Αυτό προφανώ ε, είναι βαρύ φορτίο για τι ε, εποπτικέ, για τι αρχές διαχείριση. Έχει γίνει πρόοδο, αλλά η προοδό η είναι μάλλον μετριοπαθή, δεν είναι και επαναστατική. Είναι το αποτέλεσμα των, ε, της νομοθεσίας των οδηγιών που δίνουν κατευθυντήριες γραμμές και κάποιες αρχές για την εποπτεία. Αλλά εδώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για εθνική ερμηνεία των γραμμών αυτών. Εμείς από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προσπαθούμε να προωθήσουμε την ομοιογένεια, αλλά και πάλι τονίζουμε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας και το περιθώριο διακριτικής ευκαιρίας που έχουν τα κρατημέλη είναι πάρα πολύ μεγάλο και άρα η δυνατότητα εφαρμογής και προώθηση της ομοιογένειας είναι πολύ δύσκολη. Τι θα κάνουμε λοιπόν στο μέλλον. Θα συνεχίσουμε στο πλαίσιο της ελάχιστης ε, ε, εναρμόνισης και στο πλαίσιο αυτό να σας πω από πλευράς μας ε, ότι η ανάθεση πιο πολλών πόρων, πόρων στην αρχή μας θα σημαίνει ότι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο γρήγοροι, πιο αποδοτικοί θα μας βοηθούσε. Κατά δεύτερον, εργαλεία όπως οι καταυστηρίες γραμμές είναι πάρα πολύ ωφέλιμα, αλλά το να έχουμε συγκεκριμένες εντολές που ορίζονται από τις συνθήκες μας δίνουν πιο δεσμευτικό χαρακτήρα. Και δίνουν πιο δεσμευτικό χαρακτήρα και στην δευτερογενή νομοθεσία. Μεγαλύτερο συντονισμό επίσης χρειαζόμαστε για να βρίσκουμε τις κοινέ αδυναμίες και σε ό,τι αφορά τα εποπτικά συμβούλια του IMS, θεωρώ ότι είναι σημαντικός ρόλος τους, μιας και τους δίνει και σημαντικό ρόλο και η νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο επίπεδο φιλοδοξία, σε δεύτερο βήμα θα πρέπει να κινηθούμε σε ένα επίπεδο η τρονία οδηγία, ξέρετε, είναι πιο πολύ βασίζεται σε αρχές. Εμείς θα θέλαμε να βασιζόμαστε σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φιλοδοξία μας. Να έχουμε δηλαδή οδηγίες οι οποίες θα έχουν πιο συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα δώσουν και πιο άμα, συγκεκριμένες ε, εξουσίες ε, στις αρχές AML στα κρατημέλη να έχουν δυνατότητα επιβολής κυρώσεων πέρα από το εποπτικό σκέλος του CRD. Και τέλος, όπως ξέρετε, πάντα υπάρχει δυνατότητα ομοιογένειας των εθνικών ε, εποπτών ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ξέρετε, δεν έχει εποπτικό χαρακτήρα η εντούλη τη Ευρωπαϊκή Αρχής Τραπεζών. Θα θέλαμε λοιπόν μεγαλύτερη ε, ομοιογένεια για να υπάρχει δυνατότητα δίωξη τέτοιων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό και με χαρά θα σας απαντήσω στις ερωτήσεις σας να επαναλάβω πόσο εκτιμώ το ότι με καλέσατε να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση για το πάρα πολύ σημαντικό σου θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα αρχίσω ευχαριστώντας σας που με προσκαλέσατε εδώ σήμερα για μια ακόμα σημαντική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πώς εμείς εφαρμόζουμε την νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Ξέρω το Κοινοβούλιο το συζητάει και είναι μια καλή ευκαιρία και για μας να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει υψηλή προτεραιότητα στο θέμα της καταπολέμησης της νομοποίησης παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Ακούσαμε και διάφορες εκθέσεις που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Ιούλιο και που δείχνουν πολύ καλά πόσο μεγάλη είναι η δέσμευσή μας προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Υπάρχουν και τα μαθήματα που έχουμε πάρει από το παρελθόν και διάφορες πρωτοβουλίες προκειμένου να εφαρμόζεται καλά η οδηγία για την καταπολέμηση νομοποίησης παράνομου χρήματος. Οι διάφορες μονάδες πληροφοριών συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία ακόμα περισσότερο. Για πρώτη φορά έχουμε συμπεριλάβει και διάφορες περιπτώσεις νέες που έχουμε εντοπίσει και έχουμε και μια πολύ πρακτική έκθεση για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον με μητρώα τα οποία, οποία καταγράφονται οι διάφορες επικράτειες και έχει να κάνει με τους Πραγματικού δικαιούχου το Μητρό αυτό πραγματικών δικαιούχων. Θα ήθελα να αναφερθώ στου κινδύνους, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, και για κάποιε χώρε που θεωρούνται ότι είναι κινδύνου. Όπως γνωρίζετε, το Μάρτιο που μα πέρασε, το Συμβούλιο απέρριψε μια κατεξοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με κατάλογο με χώρες κινδύνου. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά για διαφορετικού λόγου. Επαναλαμβάνω εδώ τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει αποτελέσματα με, μια, με έναν ενημερωμένο κατάλογο χωρών βάσει των νομικών υποχρώσεων που έχουμε και απορρέουν από την Οδηγία για την Καταπολέμηση Νομοποίησης Παρόνομου χρηματο. Τι έγινε λοιπόν έκτοτε από το Μάρτιο και μετά. Πρώτα απ' όλα υπήρξε ένα σημαντικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου που λάβαμε πάρα πολύ σοβαρά και βασιστήκαμε σε αυτό για να προσπαθήσουμε την άνοιξη και το καλοκαίρι να λάβουμε υπόψη μας τις ε, απόψεις που εκφράζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να πετύχουμε συνένεση μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων για τη διαδικασία προκειμένου να αποφύγουμε τη μία το Συμβούλιο, την άλλη το Κοινοβούλιο να απορρίπτουν τον κατάλογο αυτό επικίνδυνων χωρών που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για μας. Το πρώτο μου μήνυμα είναι ότι η επόμενη κατεξοδότηση πράξη θα ακολουθήσει μια αυτόνομη διαδικασία για την προστασία οικονομικών συμφερόντων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο σας, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτονομία σε αυτό τον κατάλογο. Τώρα τα κριτήρια της οδηγίας ξέρετε ότι ξεπερνούν τα κριτήρια τα οποία ακολουθεί η Task Force για την προστασία των οικονομικών ε, συμφερόντων και που αναφέρεται κυρίως ε, στο θέμα της διαφάνειας για τους πραγματικούς δικαιούχους. Στην πραγματικότητα δηλαδή οι τρίτες χώρες που έχουν ε, κάποιες αδυναμίες βάσει των ευρωπαϊκών κριτήριων θα μπαίνουν στον κατάλογό μας ακόμα και αν δεν είναι στον κατάλογο της Task Force. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θέλει να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα, λαμβάνοντα υπόψη διάφορες πηγές. Θα χρησιμοποιήσουμε και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Task Force, αλλά και τις πληροφορίες που συλλέγουμε από αποστολές που έχουμε κάνει σε διάφορες χώρες που υπάρχουν στο μητρό μας ή από επισκέψεις που έχουν κάνει εκεί, Europol, Eurojust κλπ. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, τι σχεδιάζουμε να κάνουμε. Να ξαναδούμε την μεθοδολογία που εγκρίναμε τον Ιούνιο. Και εδώ θα αναφέρω τα κύρια στοιχεία που έχουμε υπόψη μας. Πρώτον, θέλουμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες προκειμένου να τους δώσουμε κίνητρα να έχουν ένα καλό καθεστώς, καλές προδιαγραφές για την αποφυγή παράνομων τέτοιων δραστηριοτήτων. Και το συζητάμε μαζί τους πριν τις βάλουμε στον κατάλογό μας. Οπότε είπαμε ότι θα δούμε κάπως την μεθοδολογία μας και θα κάνουμε μια προκαταρτική εκτίμηση και αξιολόγηση των αδυναμιών τέτοιων χωρών. Οπότε οι τρίτες χώρες θα είναι ενήμερες και θα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ε, που βρίσκεται η διαδικασία που τις αφορά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για αυτές τις τρίτες χώρες προκειμένου να λαμβάνουν δράση και να καλύπτουν τις αδυναμίες τους. Και αυτό θα είναι το δεύτερο βήμα στη διαδικασία μας δηλαδή να βοηθάμε τις χώρες οι οποίες αναλαμβάνουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις και θα τις βοηθήσουμε συγκεκριμένα κριτήρια, με συγκεκριμένα προγράμματα δράσης για να προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις τους. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έπειτα, ε, είναι σημαντική συζήτηση με τις χώρες για να δούμε τι θέλουν. Υπάρχουν χώρε οι οποίε είναι διαδεθμένε να συνεργαστούν μαζί μας και σε εκείνες δίνουμε χρόνο στη διάθεσή τους. Χρόνο για να προχωρήσουν σε φιλόδοξες μεταρρυθμίσει και να τηρήσουν τα κριτήριά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εννοείται ότι θα παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία με επισκέψεις στη χώρα και εννοείται ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα ενημερώνονται πλήρω για όλα αυτά. Επίσης στη ε, διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και συντονισμός με τις χώρες μέλη, να ενημερώνονται και γι' αυτό και η διαδικασία θέλουμε να διέπεται από πλήρη διαφάνεια. Αυτό λοιπόν είναι το θετικό σενάριο. Ε, μάλλον το ε, κακό σενάριο σε περίπτωση που δεν τηρήσουν τα κριτήρια οι χώρες αυτές. Σε αυτή την περίπτωση θα μπουν στον κατάλογό μας ε, ως υπόχρεες οντότητες. Χώρες οι οποίες επίσης δεν συνεργάζονται, οπότε δεν τηρούν τα κριτήρια, εκείνες δεν θα έχουν καν ε, περίοδο χάριτος. Το ίδιο ισχύει και για τρίτες χώρες. Αλλά είναι σε κάπως διαφορετική κατάσταση γιατί εκεί ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος και η απειλή. Σε μερικές περιπτώσεις δεν υπάρχει κυβέρνηση ή ένα μέρος της επικράτειας δεν ελέγχεται, οπότε δεν υπάρχουν και προκτικές να τηρήσουν τίποτα κριτήρια εκείνες. Πάντως πιστεύουμε ότι μια τέτοια νέα προσέγγιση από τη δικιά μας την πλευρά θα διασφαλίσει την προστασία του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος όπως θέλουμε. Άπαξ και οι χώρες έχουν μπει στον κατάλογο και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Τι γίνεται μετά. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι άπαξ και μια χώρα μπει στον κατάλογο και πάλι δεν την αφήνουμε μόνη της. Συνεχίζεται ο διάλογος με αυτές τις χώρες και θα προσφέρουμε όσο μπορούμε περισσότερο τεχνική αρρωγή για να διορθεί η κατάσταση γιατί αυτός ο κατάλογος, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί ένα μέσο, εργαλείο, δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Θέλω να επαναλάβω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη σχέση ανάμεσα στην ε, διαδικασία που λαμβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την FATF, την Task Force. Εδώ να ξέρετε ότι διάφοροι ήρθαν σε επαφή μαζί μας να μας πούνε ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί υπάρχουν και τα δύο και τι συμβαίνει. Λοιπόν, εμείς θα διατηρήσουμε την προσέγγιση μας που λέει ότι άπαξ και μια χώρα βρίσκεται στον κατάλογο της FATF, θεωρείται υψηλού κινδύνου και έτσι τη θεωρούμε και εμείς. Επίσης όμως θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι άπαξ και η FATF αφαιρέσει από το δικό της τον κατάλογο μια χώρα δεν σημαίνει ότι αυτόματα αφαιρείται και από τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αφαίρεση από το δικό μας κατάλογο γίνεται μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιθεωρήσει και έχει διαπιστώσει ότι όντως τα δικά μας κριτήρια τηρούνται πλήρως. Θα σταματήσω εδώ νομίζω. Απλώς θέλω να επιβεβαιώσω και πάλι ότι για μας η καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση είναι θέματα που αντιμετωπίζουμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Προσπάθησα εδώ να σκεγγραφίσω λιγάκι μέσα σε λίγα λεφτά τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει για να έχουμε στη διάθεσή μας ένα αποτελεσματικό μέσο. Θα σταματήσω εδώ την εισαγωγή μου και από εδώ και πέρα είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ήδη όμω από τώρα θέλω να σα πω ότι έχουμε μια τεχνικού επίπεδου συνάντηση την επόμενη εβδομάδα για την καταπολέμηση νομιμοποίηση παράνομου χρήματο και εκεί θα συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες, ώστε να ξέρετε με κάθε λεπτομέρεια πώς έχουν τα πράγματα και ότι συνεχίζεται η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε τώρα στις ε, ερωταπαντήσεις. Ε, πέντε λεπτά ε, για τον καθένα προβλέπονται. Στο τέλος θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια διαδικασία catch the eye και παρακαλώ να με διορθώνετε αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Καταρχήν, ε, εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος ε, Κάζα. Ε, αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική Νομίζω όλοι συμφωνούμε με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια μπορέσαμε πράγματι να ε, ενισχύσουμε τους, ε, την νομοθεσία σε αυτό τον τομέα και αν η νομοθεσία και οι νόμοι εφαρμόζονται σωστά, πράγματι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ε, την νομιμοποίηση, από παράνομες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η κείμενη νομοθεσία. Και γιατί το αναφέρω αυτό, διότι ε, τα τελευταία χρόνια ε, είδαμε να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες ε, πολλοί οργανισμοί αφέθηκαν στην τύχη τους, δεν έγινε απολύτως τίποτα και νομίζω ήταν σαφές ότι είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις διεθνούς διαφθοράς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Θα έχετε ακούσει παραδείγματος χάρη ε, για την ε, τράπεζα αυτή που ε, λειτουργούσε στην Μάλτα και η άδεια της τράπεζας αφαιρέθηκε μετά από ένα χρόνο. Δηλαδή για ένα ολόκληρο χρόνο συνέχισε τις τραπεζικές συναλλαγές χωρίς καμία απολύτως συνέπεια. Το κοινοβούλιο αυτό, φαντάζομαι θα θυμάστε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξέφρασε την ανησυχία του ε, σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος ε, που γινόταν από αυτή την τράπεζα. Θα μπορούσα να αναφέρω και πολλές άλλες περιπτώσεις ε, κατά τις οποίες οι εθνικές αλλά και οι ευρωπαϊκές αρχές δραστηριοποιήθηκαν μόνο μετά ε, τον εντοπισμό των υπετίων από πλευράς όμως ε, Αμερικανικών αρχών. Εμείς δηλαδή στην Ευρώπη δραστηριοποιηθήκαμε μόνο αφού είχε ε, ξεκινήσει η υπόθεση από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και γι' αυτό λοιπόν διερωτώμε ποιε ποιες είναι οι δυνατότητες μας ως ευρωπαϊκοί και εθνικοί θεσμοί στο να λάβουμε δράση κατά των τέτοιων δραστηριοτήτων ε, τη στιγμή που οι Ηνωμένε Πολιτείε κατά κύριο λόγο είναι εκείνες οι οποίες δραστηριοποιούνται περισσότερο από όλους. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τώρα έχει περισσότερες αρμοδιότητες για να αντιμετωπίσει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτή είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, αλλά διρωτώ με άραγε αρκεί αυτό. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, γιατί φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε και πάλι νέα προβλήματα ε, όπου χρηματοψηφιακά ιδρύματα θα εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες ε, και θα προστατεύονται από ε, αυτούς που έχουν εξουσία. Δεν διευκρινίσατε όμως ε, προς ποιον απευθύνει την ερώτηση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Ε, να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι κατά κύριο λόγο επισημάνατε το γεγονός ότι είχαμε δυνατότητα να αντιδράσουμε σε κάποιες περιπτώσεις και έτσι υπήρξε και μία σύγκριση ανάμεσα στο τι κάνουμε εμείς και το τι κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα ε, των δράσεων το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών ε, κατά κύριο λόγο είναι σύστημα προληπτικό. Ενώ εμείς είμαι ένα σύστημα που λειτουργεί εκ των υστέρων. Να σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Ε, κυρίως ε, ως αρμόδια αρχή, εποπτική, αυτό που κάνουμε εμείς είναι κατά κύριο λόγο την ανάλυση κινδύνων ε, προσπαθούμε να ε, εντοπίσουμε τους σπόρους, αλλά ε, θέλω να σας πω ότι δεν είναι αλήθεια ότι η κίνδυνη είναι μηδενική. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιπτώσεις, η δική μας η δουλειά είναι κατά πόσον η αρμόδια αρχή ζήτησε από τις τράπεζες να ακολουθήσουν σωστή ανάλυση διαχείρισης ε, κινδύνου. Και αυτό που μας ενδιαφέρει ε, είναι και το τι ακριβώς προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία. Εκτός από την περίπτωση της ε, Μάλτας που αναφέρατε, πράγματι υπήρχε περίπτωση παραβίασης ενωσιακού δικαίου και οι αρχές της Μάλτας πρότειναν μέτρα πάρα πολύ χρήσιμα. Η δική μας η δυνατότητα να εντοπίσουμε τέτοιου είδους ε, αρχές, ε, οι δικές μας δυνατότητες δεν υφίστανται και κατά κύριο λόγο η δική μας η δουλειά είναι να ρωτάμε, όπως σας είπα, να εντοπίζουμε κατά πόσον οι αρμόδια έχουν προβεί σε ανάλυση διαχείριση κινδύνου. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι η δυνατότητα να εντοπίζεται κάποιος ε, σημαίνει απαραίτητα ότι το σύστημα είναι αποτελεσματικό. Σημασία έχει να υπάρχει συνεργασία έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εντοπίζονται ε, οι περιπτώσεις. Είπα στην αρχική μου παρέμβαση ότι ε, προσπαθούμε να έχουμε ομάδες ανθρώπων που ασχολούνται σε συγκεκριμένες τράπεζες με την αντιμετώπιση ε, του ε, ξεπλήματος. Όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου, θέλω να σας πω ότι κάναμε πάρα πολλά, αποκινούμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να έχουμε αυστηρότερη νομοθεσία, αλλά ε, τελικά δεν την κάνει κανείς νομοθεσία αν δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Εξάλλου, είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βλέπει πώς λειτουργούν ε, όλα αυτά ε, σωστό είναι να είναι ε, σωστές οι ε, νομοθετικές διατάξεις επίπεδο θεωρίας, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται και στην ε, πράξη συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο της Ευρώπης, στέλνουμε σε όλες τις χώρες ομάδες για να δουν κατά πόσο υπάρχει αρκετή συνεργασία, αν υπάρχει εποπτεία. Όταν υπήρξε μία περίπτωση ε, παραβίασης του νοσιακού δικαίου, το ανέφερε αυτό προλαλή ε, ε, και η περίπτωση αφορούσε και τη Μάλτα, είδαμε τότε ότι δρομολογήθηκαν πάρα πολλές εξελίξεις και στο τέλος ε, ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ε, δραστηριότητες για να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία στις διάφορες χώρες. Τώρα συνεργαζόμαστε με κράτη-μέλη ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της. Θα ήθελα να παρακαλώ, παρακαλέσω τους αδέλφους ε, να είναι πιο σύντομες ερωτήσεις τους για να υπάρχει χρόνος για ε, πιο ε, περιεκτικές απαντήσεις. Ο κύριος Τάνκ. Ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα για την αλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι εδώ στην αίθουσα πιστεύουν ότι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εισόδων από εγκληματικέ ενέργειες είναι σημαντικό. Το θέμα είναι πώ θα συμφωνήσουμε σε θέματα εφαρμογή στη φάση αυτή σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τράπεζες οι οποίες δεν ε, καταφέρουν, καταφέρνουν να ανταποκριθούν στα πρότυπα και στις προδιαγραφές που έχουμε θέσει. Και το παράδειγμα είναι η ING. Η ING η οποία ε, δήλωσε ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν σωστό ευρωπαϊκό συντονισμό. Να ξεκινήσω εδώ, γιατί μία πτυχή είναι ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των IFIU και των ε, αρχών εφαρμογή του νόμου είναι προβληματικό. Δεν πηγαίνει τόσο καλά όσο θα έπρεπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντα υπέρ ενός ε, συστήματος ευρωπαϊκού FIU για να υπάρχει πιο αποτελεσματικό συντονισμό ε, τη συνοριακή ε, συνεργασία, τη συνοριακού συντονισμού. Μιλάμε λοιπόν για την εφαρμογή όχι μόνο στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο εξωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και έχουμε ένα κατάλογο, μάλλον θα ήταν πολύ απαραίτητο να έχουμε ένα κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου για να καταπολεμήσουμε τις ε, απειλές αυτές και είναι πραγματικά κρίσιμο για μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια διαδικασία για πιο αυστηρά κριτήρια από αυτά που ζητούνται από το FTF, κυρίως ό,τι αφορά τα θέματα διαφάνειας και των ε, ε, δικαιούχων. Και να ρωτήσω λοιπόν, πιστεύετε ότι αυτά τα στοιχεία θα είναι ανοιχτά για δημόσια, εμ, δημόσιο έλεγχο από το κοινό, γιατί αυτό θεωρώ ότι θα καθορίσει την αξιοπιστία. Και επίσης τι γίνεται ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι γίνεται με τα δημόσια μητρώα για θέματα της κυδεκτησίας. Ευχαριστώ πολύ και αν καταλαβαίνω σωστά το ερώτημα ήταν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πω δύο λόγια καταρχάς για το θέμα της αξιοπιστίας ό,τι αφορά θέματα εφαρμογής. Όντως, το καλοκαίρι και το αναφέραμε και στην έκθεση. Κάναμε μια εσβάθος ανάλυση του τι πήγε καλά και τι πήγε στραβά. Εδώ θα βρείτε λοιπόν σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εφαρμογή τι έγινε από τις διάφορες αρχές. Και εδώ θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Η έκθεσή μας το δηλώνει αυτό με σαφήνεια. Επίσης, συμφωνώ μαζί σας ότι σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των FIU και των άλλων φορέων, ε, παράδειγμα αρχές επιβολής του νόμου, αλλά και FIU σε άλλα κρατημέλη, θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Κάναμε ένα πρώτο βήμα με το προηγούμενο κοινοβούλιο για την ε, νέα αυτή διάσταση. Αλλά πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα σημείο που μας απασχολεί. Για τις ε, χώρες υψηλού κινδύνου τώρα. Και για τα benchmarks, για τα σχέδια δράσης. Συμφωνούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τη δέσμευση του Ευρωπαίου νομοθέτη. Κατά πόσο αυτά τα benchmarks θα πρέπει να είναι δημόσια, θα πρέπει να το σκεφτούμε. Αλλά σας ευχαριστώ που το θέσατε ως ερώτημα. Γιατί ενδεχομένω να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, οπότε θα πρέπει να δούμε τα υπέρ Να δούμε τι γίνεται και στο FRTF. Δεν σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει να αντιγράψουμε ακριβώς την διαδικασία, αλλά το σημειώνω ότι το θέσατε για το θέμα των δικαιούχων. Ε, είμαστε στην ίδια γραμμή. Πιστεύουμε ότι το σύστημα αυτό ενδεχομένω να είναι το πιο φιλόδοξο σε ό,τι αφορά και την καταχώρησή τους. Στην παρούσα φάση, να σας πω ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε στο 30F αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο πολύ σύστημα σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους και μητρώα. Αυτό θα συνεχίσουμε να το προωθούμε. Κάποιες χώρες είναι λίγο πιο ανοιχτέ από ό,τι άλλες, αλλά θα πρέπει να το τονίσουμε και να το θέσουμε και στους ε, διεθνείς εταίρους μας. Είναι βασικό το θέμα αυτό. Δεν πρόκειται να το καταφέρουμε μέσα σε μία νύχτα, αλλά θα πρέπει να καλέσουμε και τις άλλες ε, αρχές ε, να κινηθούν προ την κατεύθυνση αυτή, να κάνουν το σύστημά του πιο διαφανές. Ε, ο κύριος Λουίδη Καρικάνα από το Ρενιού τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η καταπολέμηση νομοποίησης παράνομου χρήματος είναι όπως αυτές οι χαρακτηριστικές ε, περιπτώσεις που κάνουν οι θεσμοί τη δουλειά χωρίς πάντα τα αποτελέσματα γιατί δεν διαθέτουν τα σωστά μέσα, όπως είπε και ο κύριος Κάμπα για την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Είναι σαν να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε να κάνουμε. Και γιατί, γιατί οι χώρες κλείνουν τα μάτια και τελικά το σύστημα είναι τόσο δυνατό όσο είναι ο πιο αδύναμος κρίκος του κανείς δεν κάνει τη δουλειά του τελικά. Και τελικά φτάνουμε στο ότι, όπως λέει και ο κύριος Κάμπα, δεν έχουμε πραγματική εναρμόνιση. Θέλω λοιπόν τρεις ερωτήσεις να υποβάλω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, ο δρόμος που ακολουθούμε τώρα, που είναι οδηγίες και οι χώρες αποφασίζουν για την συμμόρφωση, πότε τελικά γίνεται ή όχι, δεν φαίνεται να λειτουργεί γιατί τα κίνητρα δεν είναι σωστά για τις χώρες. Οπότε μήπως θα μπορούσαμε να πάμε σε κανονισμό που διασφαλίζει την ε, εναρμόνιση με κυρώσεις κλπ. Δεύτερον, ο κύριος Κάμπα αναφέρθηκε στο Συμβούλιο Εποπτών. Θα ήταν λογικό να υπάρχει ένας θεσμός που να μπορούν μέσα σε αυτό να συναντιόνται οι υπεύθυνοι όπως γίνεται στο Ευρωπαϊκό Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Τι εμπόδια υπάρχουν για να ελοπιθεί κάτι τέτοιο. Και τέλος, στην Επιτροπή πάντα. Ποιο είναι το εμπόδιο και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να έχει τα μέσα που χρειάζεται και τους πόρους που χρειάζεται, προσωπικό, χρήματα. Γιατί δεν μπορεί να υποσχόμαστε στους πολίτες ότι θα κάνουμε μια δουλειά για την οποία δεν πρικοδοτούμε τους αρμόδιους επαρκώς. Και θέλω να πω στον κύριο Κάμπο ότι τον στηρίζουμε. Εδώ είμαστε όλοι οι ευρωβουλευτές και διαβεβαιώνουμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε το θέμα αυτό και γι' αυτό και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να μπορέσει να έχει τα μέσα που χρειάζεται. Κύριε Κάμπα, έχετε μεγάλη πρόκληση μπροστά σας για την καταπολέμηση παράνομου χρήματος. Το ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανωνυμία. Εσείς πώς θέλετε να αντιμετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις. Ωραία, Ευρωπαϊκή Επίτροπη πρώτα. Ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση τι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για την καταπολέμηση νομιμοποίηση παράνομου χρήματος. Πρέπει κανείς να έχει ανοιχτό μυαλό. Έχουμε την οδηγία, έχουμε προχωρήσει ήδη πολύ. Υπάρχουν βελτιώσεις, δεν ξέρουμε βέβαια πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Και πρέπει επίσης να κρίνουμε, να εκτιμήσουμε τι έχει λειτουργήσει καλά στην οδηγία, τι όχι. Αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι θα το δούμε, αλλά χρειαζόμαστε πρώτα περισσότερη ανάλυση για να δούμε τι γίνεται καλά, τι όχι, τι θα μπορούσε να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή γιατί πράγμα πρέπει να αφήσουμε περισσότερη ευελιξία στις χώρες μέλη. Πάντως σίγουρα είναι κάτι που το εξετάζουμε και το παίρνει πολύ σοβαρά η Επιτροπή. Για το Συμβούλιο Εποπτών. Για μας, καλά, ο τίτλος δεν έχει και πολύ σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι όντω να μπορούν να βρίσκονται άνθρωποι μεταξύ τους. Γιατί το έχουμε δει και εμείς, ότι οι άνθρωποι δουλεύουν ε, σε διαφορετικούς δρόμους, αλλά για να πετύχουν τον ίδιο στόχο τελικά. Οπότε έχουμε την αίσθηση ότι μερικές φορές λείπει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, να θέλουν οι μεν να μοιράζονται πληροφορίες με τους δε, χωρίς να νιώθουν ότι υποχωρούν σε κάτι. Το Συμβούλιο Εποπτών θα μπορούσε να είναι μια λύση, χωρίς να έχει σημασία το πώς θα λέγεται. Αρκεί να υπάρχει συνεργασία. Για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πρέπει να είμαι κάπως προσεκτική, γιατί εγώ είμαι στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, οπότε δεν ασχολούμαστε με την EBA. Αυτό όμως που μπορώ πράγματι να πω είναι ότι οι πόροι για την καταπολέμηση νομοποίησης παράνομου χρήματος είναι ε, σημαντικοί. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, αρκετό προσωπικό που δουλεύει. Πιστεύουμε και εμείς δηλαδή ότι ναι, πρέπει να υπάρχουν αρκετοί πόροι. Καλώς, ευχαριστούμε. Κύριο Κάμπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά τους πόρους, ξέρετε, συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Διεύθυνση δικαιοσύνη Είναι αλήθεια ότι μας έχει στηρίξει, έχει ζητήσει να αυξηθούν οι πόροι για όλες τις χώρες όσον αφορά το AML, την καταπολέμηση δηλαδή νομοποίηση παράνομου χρήματος. Τρεις έχουμε που δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα από τον Απρίλιο. Για ένα χρόνο θα είναι αυτό. Θα βοηθούσε πράγματι να έχουμε περισσότερους Όσον αφορά ε, τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, έχει στείλει προειδοποίηση η, EBA σχετικά με αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο τα κρυπτονομίσματα, εμείς το λέμε πιο πολύ κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, γιατί είναι κάτι παραπάνω. Και έχουμε ειδοποίηση για τους κινδύνους. Και είναι και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Πάντως, το έχουμε υπόψη μας. Εμείς είμαστε μια τραπεζική αρχή. Πάντως, το νέο με την εξέλιξη αυτή είναι ακριβώς ότι επειδή δεν μπαίνει στο σύστημα, δεν είναι σίγουρο ότι η νομοθεσία ε, το πιάνει αυτό το φαινόμενο. Γιατί μπορεί να είναι επενδύσεις, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Λοιπόν, για το ηλεκτρονικό χρήμα έχουμε το σχετικό μητρίο, μητρό, αλλά υπάρχει πράγματι κάποιο κενό εδώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου των Πρασίνων, ο Σβέν και Γκόλτ. Παρακαλώ τους ομιλητές να είναι σύντομοι στις ερωτήσεις τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ε, καταγράψαμε όλες τις δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πριν από το καλοκαίρι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό ε, και ακούσαμε και τη νέα μέθοδο που προτείνεται. Βεβαίως είναι ντροπή το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν ενέκριναν αυτόν τον μαύρο κατάλογο και τώρα έχουμε μια νέα μέθοδο ε, σχετικά με τη μεθοδολογία. Όσον αφορά τη μεθοδολογία σας, κυρία Σρούντερ, έχω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Συγκρίνοντας αυτή τη μεθοδολογία με τον μαύρο κατάλογο περί φορολογίας, υπάρχει ένας γκρίζος ε, κατάλογος, όπου κάποιες χώρες είναι ύποπτες, εξετάζονται και περιμένουμε να γίνουν ε, κάποιες κινήσεις. Αυτά για τη φορολογία. Εσείς ε, στη δική σας την πρόταση, γιατί δεν έχετε αυτή τη γκρίζα λίστα Τώρα, κάτι άλλο. Υπάρχει ε, και ένα, μια καταληκτική ημερομηνία 12 μηνών για κάθε χώρα. Ε, αρχικά, νομίζω, θέλετε 6 μήνες. Άρα, δηλαδή, υπάρχει κάποιος κίνδυνος από κάποια τρίτη χώρα. Και τι κάνουμε, περιμένουμε 12 μήνες και δεν κάνουμε τίποτα. Και κάτι άλλο, όταν βλέπετε να υπάρχουν προβλήματα και τα αναλύετε, ε, αν δεν υπάρξει αυτός ο κατάλογος ε, με κατεξοδότηση πράξης, μπορεί να περάσουν μέχρι και 18 μήνες. Και από τότε που ε, γίνεται η ανάλυση μέχρι να ληφθούν μέτρα, περνάνε 18 μήνες. Αυτό όμω είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για λόγους ασφαλείας. Και όσον αφορά το FATF, εάν ε, κάνουν ανάλυση, δημοσιεύουν μία έκθεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει ανοιχτή και διαφανή διακυβέρνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν το γεγονός ότι οι δικές σας οι εκθέσεις αξιολόγησης δεν πρόκειται να δημοσιευτούν. Πρέπει να δημοσιεύονται οι εκθέσεις και γι' αυτό το λόγο εγώ ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόζει πιο αυστηρή μέθοδο, ακριβώς όπως το έχουμε ζητήσει και να μην ενδίδεται στην πίεση των κρατών μελών που είναι όσον αφορά την ε, καταγραφή σε καταλόγους τρίτες χώρες να υπάρχει έτσι μια γενικότερη χαλαρότητα. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ε, ερωτήσεις. Ε, τα σημείωσα σας είπατε και θα τα κοιτάξουμε και αργότερα. Δεν μπορώ να σας πω α, ακριβώς, θα να σας δώσω όλες τις απαντήσεις. Ε, πολύ σύντομα να σας πω το εξής. Το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος ε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα νομικής φύσεως θέμα, γιατί ο πραγματικός κατάλογος θα πρέπει να γίνει ε, στο άρθρο 9, ε, όπου να υπάρχει μια απόφαση σχετικά με τα στρατηγικής φύσεως προβλήματα. Κύριε Γκίκολτ, αν κατάλαβα καλά, αυτό τον βλέπετε περισσότερο ως πολιτικό και όχι ως νομικό κατάλογο. Εγώ ήμουν απόλυτα σαφή, λέει ο κύριο Γκίκολτ. Κοιτάξτε, στα φορολογικά, όταν μια χώρα εντοπιστεί ότι δημιουργεί προβλήματα και περιμένουμε να εφαρμοστεί η νομοθεσία, σε αυτό το χρονικό διάστημα η χώρα μπαίνει σε γκρίζα λίστα. Εσεί δεν προτείνετε γκρίζα λίστα, γιατί ε, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ε, οποτεδήποτε πιστεύουμε ότι μια χώρα δημιουργεί προβλήματα. Σβέν, αν θέλεις και αργότερα μπορείς να ρωτήσεις. Κοιτάξτε, ε, δεν μπορώ να σας πω σήμερα ναι ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε, θα δούμε αν μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι, όπως έγινε και με τον ε, κατάλογο ε, για τα φορολογικά. Όσον αφορά τις καταληκτικές ημερομηνίε, ε, πράγματι δεν θα πρέπει να είναι πολύ μακριά ούτε και πολύ κοντά, να είναι ρεαλιστική καταληκτική ημερομηνία που θα επιτρέπει σε μια χώρα να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ε, νομοθετικές αλλαγές, κοινοβουλευτικές διαδικασίες ε, και δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να έχουμε μια ημερομηνία που να μην μπορεί να τηρηθεί. Επίσης, να μην είναι η καταληκτική ημερία, ε, ημερομηνία πολύ μακριά για να πιστεύουν όλοι ότι έχουν ε, πάρα πολύ χρόνο. Όσον αφορά στις εκθέσεις ε, και πώς θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Όπως είπα στην εισαγωγική μου παρατήρηση, υπάρχει μία δέσμευση ότι σε όλη τη διαδικασία το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται θα ενημερώνεστε σχετικά με τις αξιολογήσεις μας και θα μπορείτε και να τις βλέπετε. Ένα άλλο ερώτημα που ε, τέθηκε αφορά τη δημοσιοποίηση προς την κοινή γνώμη, προς τα έξω. Το σημείωσα και όπως σας είπα θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τι έγινε στο FATF. Ε, εδώ βέβαια είναι λιγάκι διαφορετικό το θέμα αλλά εν πάση περιπτώσει ε, θα δούμε ε, σε τελική ανάλυση τι προκύπτει, αλλά τα έχω σημειώσει όλα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ, Μπέρκ, από το ID. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα με την Europol, περίπου 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ είναι από παράνομες προσόδους. Και αυτό ανέρχεται περίπου στο σύνορο του Ευρωπαϊκού Προεπιλογισμού. Τον Ιούλιο του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία δήλωση σύμφωνα με την οποία θεωρεί ότι η καταπολέμηση των παράνομων αυτών προσόδων ε, ήταν πιο αποτελεσματική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα με οδηγία και όχι σε εθνικά επίπεδο. Η πέμπτη οδηγία για το ξέπλυμα χρήματο θεωρήθηκε εμ, ανεπαρκής ε, για την επιτευχή των στόχων που είχε θέσει. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, θεωρείται ότι έλαβε περαιπάνω, μάλλον αρμοδιότητες ε, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των με Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ότι και οι αρμόδιοτητες αυτές είναι ανεπαρκείς. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσει να σας κάνω. Τι περαιτέρω αρμοδιότητες πιστεύετε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εναποθέσουν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τι συγκεκριμένα προβλήματα θα συνεπαγόταν ε, μια τέτοια κοινοτική διαμόρφωση των ελέγχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι προβλήματα επέλυε. Κατά δεύτερον, συμφωνείτε με εκείνους που θεωρούν ότι ήδη έχει αποτύχει αυτή η πέμπτη οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος, προτού καν ε, εφαρμοστεί στο ε, πλήρες από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρώτη ερώτησή σας ε, να σας πω Νομίζω ότι δεν θα είναι σωστός τρόπος να αφαιρεθούν αρμοδιότητες και να μπουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτού διαμορφωθεί μια σαφής εικόνα για το τι κάνει ποιος και ποιος θα μπορούσε να κάνει τι με καλύτερο τρόπο, με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στην έκθεση, σαν τέλη Ιουλίου, θεωρώ ότι δώσαμε μια πολύ καλή εικόνα των ε, αδυναμιών που υφίστανται σε ό,τι αφορά τις αρχές επιτόπου. Και εδώ θα πρέπει να εργαστούμε παραπέρα, παρατέρω, για να ξέρουμε που βρισκόμαστε πρωτού. Ε, πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε ευρωπαϊκές λύσεις. Είναι μία μόνο εναλλακτική, η οποία ενδεχομένω να αντίκρινεται ενδεχομένω και όχι. Αλλά χρειάζεται περισσότερη ανάλυση και από εμά και από όσου ασχολούνται με το θέμα αυτό. Για την δεύτερη ερώτηση, για την ε, οδηγία. Όντω, υπάρχει η καταληκτική ημερομηνία για την ε, υλοποίηση, την εφαρμογή τη οδηγία. Ιανουάριο του 2020. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όπω κάναμε και με τι άλλε οδηγίε, ελέγχουμε πάρα πολύ προσεκτικά κατά πόσο τα κρατημέλη έχουν ε, εφαρμόσει όλε τι νομικέ προδιαγραφέ οι οποίε προβλέπονται όχι μόνο σε ό,τι αφορά το θέμα των δικαιούχων, και των δικαιωμάτων πρόσβασης. Επί τη βάση αυτή, θα συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας για να δούμε κατά πόσο χρειάζεται περαιτέρω εργασία. Εργαζόμαστε λοιπόν με ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μα, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι σήμερα είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να αποφανθούμε. Τώρα από το ECR δεν βλέπω εδώ τον κύριο Ράπη. Αντικαθιστά κάποιο ε, τον κύριο Ράπη από το ECR. Θέλει να πάρει το λόγο. Αν όχι, ο κ. Παπαντεμούλης από την ΚΟΥ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Κάμπα, νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζουν τις προσπάθειές σας, αλλά και από ό,τι άκουσα μέχρι τώρα από ε, τους προηγηθέντες ομιλητές, κανείς μας δεν είναι ικανοποιημένος από την αποτελεσματικότητα που έχουμε μέχρι τώρα δείξει στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Γιατί είναι ένα κομμάτι του οικονομικού εγκλήματος η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Και αυτό είναι ολοφάνερο, χωρίς να είναι κανείς ειδικό, όταν μερικές δεκάδες ερευνητών δημοσιογράφων ανακαλύπτουν σκάνδαλα και φέρνουν στη δημοσιότητα σκάνδαλα νομιμοποίηση εσόδων από ξέπλυμα μαύρου χρήματος και από εγκληματικές δραστηριότητες που δεν μπορούν να τα ανακαλύψουν και να τα καταπολεμήσουν οι εθνικές αρχές, οι ευρωπαϊκές αρχές, αυτό σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Και επειδή τέθηκαν τα θέματα, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και την εκπρόσωπο της Κομισιόν και τον κύριο Κάμπα, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει για να ανεβάσουμε την αποτελεσματικότητα και των εθνικών αρχών και των ευρωπαϊκών αρχών. Τι πρέπει να αλλάξει στην νομοθεσία, τι πρέπει να ενισχυθεί σε πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς, πόσο πρέπει και πώς να προχωρήσει η συνεργασία των εθνικών κρατών με τα κράτη-μέλη και πώς θα μπορέσουμε να παρακάμψουμε τις αντιδράσεις ορισμένων κρατών μελών οι τα οποία κρατούν καθυστέρηση, βάζουν εμπόδια. Γιατί είναι μελανό σημείο στην προηγούμενη θητεία η άρνηση ε, του Συμβουλίου να εγκρίνει την περίφημη μαύρη λίστα. Αλλιώ, θα καθόμαστε εδώ, θα συζητάμε, θα συμφωνούμε μεταξύ μα, αλλά τα πράγματα δεν θα προχωρούν. Τι πρέπει να αλλάξει, από εσά περιμένουμε και προτάσεις και ενέργειες. For the Commission. Ο για μένα ε, το πρώτο στοιχείο που πρέπει να εξετάσουμε και εδώ επανέλθουμε στον τρόπο με τον οποίο συζητήσαμε σήμερα το πρωί είναι η ε, σωστή ενημέρωση. Να υπάρχει ένα πλαίσιο και υπάρχει ίσως αυτό, αλλά δυστυχώς δεν υλοποιείται. Πράγματι, τα κράτη-μέλη φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Ε, τα κράτη-μέλη οφείλουν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους ε, ε, όμως ε, βέβαια είναι ένα σημαντικό βήμα να δούμε τι έχει γίνει κατά το παρελθόν. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις και αυτά αφορούν όχι μόνο την νομική εφαρμογή αλλά και την πρακτική εφαρμογή. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει εν μια νυχτή, ε, χρειάζεται πόρους, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε επ' αυτού. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, πριν περάσουμε στον επόμενο γύρο, ε, πριν έχουμε μια σαφή εικόνα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει σωστή εφαρμογή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να διαδραματίσει το ρόλο της. Ε, κοιτάξτε, αυτά που ισχύουν αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικά και θέλω να σας πω ότι μεγάλη ευθύνη ε, βρίσκεται επίσης στα κράτη-μέλη. Ε, από εκεί εξαρτάται ε, το πόσο θα έχουμε σωστή εφαρμογή των νόμων για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Αυτό σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών ε, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τον έλεγχο με τα μέσα που έχουμε, αλλά είναι κοινή προσπάθεια με τα κράτη-μέλη. Περνάμε στο δεύτερο γύρο. Λιγότερο χρόνο, παρακαλώ, να μισή λεπτό ερώτηση. Μαξ Φέμπερ. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω να κάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Φεβρουάριο του φετινού έτου η Ευρωπαϊκή ε, αρχή εποπτεία ξεκίνησε, δραστη... ξεκίνησε ε, διαδικασία επί ενδεχομένω ενδεχομένως κατά τη Εστονικής και τη Δανική Τράπεζα σε, σε ύψους εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων. Και τα, το αποτέλεσμα, το πόρισμα ήταν αρκετά καθοριστικό. Ε, εντοπίστηκαν προβλήματα. Αλλά η, τα υποπτικά συμβούλια αποδυνάμωσαν αυτή την έκθεση. Και ξέρετε ότι κόρακα σκορά δεν βγάζει. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι αποτράπηκε μια αποτελεσματική διαδικασία και θεωρώ ότι υπέστη ε, βλάβη, σημεία η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Τι λοιπόν συνέπειες έχετε εσείς, ε, τι συμπεράσματα έχετε να εξαγάγετε, είσαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα πάω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσω και εγώ στα γερμανικά λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έλαβε την απόφαση αυτή και αποτελεί ανεξάρτητη αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων. Δεν ήταν καν στην αίθουσα όταν ελήφθησε η απόφαση εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει φυσικά τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και τον Ιούλιο στην έκθεσή μας που δημοσιεύτηκε αναφερθήκαμε στην ε, περίπτωση αυτή και την υπόθεση αυτή και κάναμε και περαιτέρω, ε, είχαμε περαιτέρω επικοινωνίε με τις αρχές της Εστονίας και της Δανίας. Είναι περιπτώσεις οι οποίες ε, είναι αρκετά παλιά βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να τις αποταχτούμε με σταυρωμένα χέρια. Αναμένουμε πληροφορίες από τη Δανία και από την Εστονία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ξέρετε ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάση, αλλά χρειαζόμαστε επαρκείς πληροφορίε για να έχουμε και νομικά τεκμήρια. Δεν έχει λοιπόν κλείσει αυτή η φάση, είμαστε σε φάση ανάλυσης ακόμα. Ο κύριο Κάμπα. Αν μου επιτρέψετε, την συντομία, να κάνω ένα σχόλιο ότι το Συμβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή Έλαβε, λήφθησαν κάποιες αποφάσεις λοιπόν στο Συμβούλιο. Να τις εξηγήσουμε. Καταρχάς, ότι το Συμβούλιο καλείται να κρίνει κατά πόσον ακολουθήκαν σωστέ διαδικασίε και υπήρχαν ποσοστοί πόροι στι εθνικέ αρχέ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη οδηγία. Όχι δηλαδή το τι έγινε στην τράπεζα, αλλά κατά πόσο ακολουθήθηκαν σωστέ διαδικασίε από τι εποπτικέ αρχέ. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η υπόθεση πάει πολύ καιρό που έχει λάβει η χώρα. Δεν υπήρχε η νομοθεσία, δεν υπήρχε η ίδια αρχή πρόληψης. και θεωρήσαμε ότι ήταν πιο τρέχον και πιο κατεπήγον να τεθούν υποθέσεις για υφιστάμενες περιπτώσεις που ήταν ακόμα, υποθέσεις που ήταν ακόμα σε υποεξέλιξη παρά να κοιτάξουμε παλιές ε, τέτοιες υποθέσεις. Ευχαριστούμε. Η κυρία Νίνα Γκίλ, εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Χαίρομαι που έχετε μια ισχυρή εντολή σίγουρα βοηθάει. Η ανησυχία μου όμως είναι ότι ίσως φαίνεστε, μιλήσατε για 11 ε, πλήρου απασχόληση ανθρώπου για να αντιμετωπίσετε την καταπολέμηση παράνομου χρήματος ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια τα οποία έχουν εξεπληθεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι πόροι για να μπορέσετε να βρείτε, να φτάσετε σε αυτό το παράνομο χρήμα. Φαίνεται ότι τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Πρέπει να υπάρχουν και κυρώσεις. Οπότε η ερώτησή μου είναι, θα λέγατε ότι οι τρέχουσες κυρώσεις φτάνουν, είναι αρκετά αυστηρές για να δρουν αποτρεπτικά. Γιατί ποιες θα ήταν οι καλύτερες κυρώσεις που να είναι και πιο αποτελεσματικές. Και πολύ σύντομα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπατε ότι οι χώρες ε, μέλη ε, έχουν αντίσταση προκειμένου να δεχτούν νέα σώματα. Τότε πώς θα γίνει ο συντονισμός καλύτερα μεταξύ των συνόρων. Και πώς θα μπορούσαμε να είχαμε μια πτέρυγα της Europol, αλλάζοντας ως την εντολή της. Και χθες η Κριστίν Λαγκάρτ είπε ότι όντω πρέπει να είμαστε πιο δραστικοί όσον αφορά την καταπολέμηση νομοποίησης παράνομου χρήματος. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ωραία, να αρχίσει η πρώτη επιτροπή. Ναι. ώστε θα μπορούσαμε να πετύχουμε καλύτερα το συντονισμό. και πάλι δεν υπάρχει μια λύση που να είναι καλή για όλους. Σίγουρα και εμείς έχουμε κάποιο ρόλο για να φέρουμε μαζί τους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα στο ίδιο τραπέζι να καθίσουν. Και έτσι να δούμε πού δεν έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά ο διάλογος ή ο συντονισμός. Γιατί και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Για την Europol ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπάρχουν ε, θεωρητικά πολλές δυνατότητες, αλλά είναι πολύ νωρίς πιστεύω να επικεντρωθούμε τώρα σε ένα πράγμα. Ναι, όντω η νομική βάση θα ήταν δυσκολία στην περίπτωση τη Europol γιατί είναι αστυνομική αρχή και δρά προληπτικά. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο και σήμερα η Europol μας έχει βοηθήσει ήδη με την ανάλυση και με τις ε, διάφορες ε, μονάδες χρηματοπιστητικής ε, σταθερότητας. Νομίζω ότι όντως η καλύτερη συνεργασία και η αμοιβή εμπιστοσύνη είναι τα βασικά ζητήματα. Υπάρχουν αδυναμίες πάνω στις οποίες πρέπει να δουλέψουμε. Ο κύριος Κάμπα. Ευχαριστώ κι εγώ για την ερώτηση. Δεν είναι επόπτης η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για το θέμα της καταπολέμησης, νομιμοποίησης χρήματος από παράνομες δραστηριότητες. Ε, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει η συνεργασία και η γνώση, αλλά πάνω απ' όλα η καλή υλοποίηση. Την εποπτεία όμως του θέματος την έχουν οι εθνικές αρχές. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Το αν αυτό λειτουργεί ή όχι, εντάξει, αλλά το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εμεί περισσότερο προληπτικά δρούμε. Οι κυρώσει είναι και το επίπεδό τους είναι θέμα εθνικό, των εθνικών αρχών. Ευχαριστούμε για το ο κύριος Αντρέ Κοβάρικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθαν να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Από τις απαντήσεις σας μέχρι τώρα φαίνεται να παραμένουν πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή μένουν αναπάντητα ερωτήματα. Θα επανέλθω σε αυτά που δημοσιεύσατε τον Ιούλιο, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε στο τρέχον πλαίσιο αδυναμίες. θα έπρεπε να υπάρχει μια εκτίμηση επιπτώσεων όταν πρόκειται για την εφαρμογή της τρέχουσας νομοθεσίας. Αλλά όπως είπανε και άλλοι πριν από μένα, ίσως θα ήταν καλύτερα να έχουμε ένα κανονισμό και όχι μια οδηγία όπως έχουμε τώρα. Θέλω να ξέρω λοιπόν μια τέτοια εκτίμηση αντικτύπου έχει γίνει, θα γίνει Πότε μπορούμε να περιμένουμε μια τέτοια εκτίμηση. Και αν ε, μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι, τι παίζει, τι λαμβάνετε υπόψη σας για να εκτιμήσετε το αν όντως πρέπει να αλλάξει και από οδηγία να γίνει κανονισμός. Ποια είναι τα κριτήρια. πριν προσαρμόσετε αυτά τα οποία δημοσιεύσατε τον Ιούλιο. Και πολύ σύντομα υπάρχουν δύο τομείς που αναφέρονται στα έγγραφα του Ιουλίου επικίνδυνες που είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τα λιμάνια. Θα ήθελα να μου πείτε πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι ανησυχίες σας και πώς σκέφτεστε να τις καθισχάσετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για την πρώτη τι θα ήταν καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι πρέπει να πω ότι κάθε φορά που θέλουμε κάτι να το αλλάξουμε πρέπει προηγουμένως να έχουμε εξετάσει τι λειτουργεί και πρέπει να κρατήσουμε και τι όχι. Οπότε το ίδιο θα γίνει και με την οδηγία όταν οι χώρες μέλη την ε, ενσωματώσουν και την εφαρμόσουν. Μετά θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τομείς όπου οι χώρες έχουν μια εντελώ διαφορετική προσέγγιση γιατί Όντω, η οδηγία βάζει ένα στόχο και κάποιε χώρε αποδεικνύονται ιδιαίτερα φιλόδοξε και προχωράνε πάρα πολύ, άλλε πιο διστακτικά. Τότε λοιπόν όταν θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία θα δούμε ε, πώς λειτουργεί και ανάλογα θα αποφασίσουμε. Ίσως σε μερικές περιπτώσεις να είναι καλύτερα να παραμένει κάποια ευελιξία ε, στις χώρες μέλη. Αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό τώρα. Θα γίνει η αξιολόγηση. Μια νέα επιτροπή θα δει τελικά ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Τώρα, αναφερθήκατε στην υπερεθνική αξιολόγηση κινδύνου. Και αναφερθήκατε σε κάποιους νέους τομείς Αναφερθήκατε στους ελεύθερους λιμένες και τον κίνδυνο που όντως είναι μεγάλος. Ε, και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο επίσης χρειάζεται διαφάνεια. Έχουμε δει περιπτώσεις κατά το παρελθόν. Έχουν ληφθεί κάποια και προληπτικά μέτρα προκειμένου να προχωρήσουμε και σε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σώτα Μαρκάρας από το ΕΛΚ. Αγαπητέ Πρόεδρε, δύο ερωτήσει έχω να κάνω. Μία προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία προ τον κύριο Κάμπα. Σα συγχαίρω και πάλι, κύριε Κάμπα, για την θέση σα, για τον διορισμό σα. Την πρόσφατη έκθεση σε ό,τι αφορά την ε, καταπολέμηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Τραπεζών κατά τη ε, ε, νομιμοποίηση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Είναι σαφέ για μένα ότι θα πρέπει να έχει σωστό προσωπικό και σωστή χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Και γι' αυτό λοιπόν ρωτώ το εξή. Τι είδου χρηματικέ, χρηματοοικονομικέ, ε, τι είδου πόρου ε, χρειάζεστε και τι είδου προσωπικό χρειάζεστε επιπλέον για να ανταπεξελθέτε στι νέε αυτέ αρμοδιότητε. Δώστε μας κάποια αριθμητικά στοιχεία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να θέλω να προκαταλάβω τα αποτελέσματα της ανάλυσης που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεταφοράς τέτοιων δραστηριοτήτων και εξουσιών σε μια κοινοτική υπηρεσία να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κάμπα, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Καταρχάς, ε, έχετε απόλυτο δίκιο ότι η πόροι μας είναι περιορισμένοι. Θέλουμε λοιπόν, θα ε, πάμε από 3-11 υπαλλήλου ε, του χρόνου στα θέματα αυτά, αλλά και πάλι είναι πολύ περιορισμένο το προσωπικό που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, το Κοινοβούλιο νομίζω για του χρόνο προβλέπει να προτείνει πέντε επιπλέον ε, θέσεις. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αυτό, γιατί είμαστε μικρή αρχή ε, και το θέμα είναι και πόσο γρήγορα μπορούμε να μεγαλώσουμε ως αρχή. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε και σωστά καταρτισμένα άτομα δεν μπορούμε ξαφνικά να προσθέσουμε 400 άτομα στο προσωπικό μας. Όσο θα προχωράμε θα έχουμε πιο πολλές ε, ανάγκες προφανώς, αλλά εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάρα, το ερώτημα που θέσατε δεν είναι απλό. Είναι και πολύ επίκαιρο, ωστόσο, γιατί συχνά ε, στρεφόμαστε προς τον τραπεζικό κλάδο σε ό,τι αφορά θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Τα πράγματα σε γενικέ γραμμέ ε, είναι σαφή στο χρηματοοικονομικό κλάδο, στο μη χρηματοοικονομικό κλάδο, όμω τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα, δεν υπάρχουν, είναι πολύ πιο μεγάλη ποικιλία. Έχουμε πολλού τομεί που μπορεί να γίνει ενδεχομένω ξέπλυμα χρήματο, αλλά διαφέρουν οι κανόνε. Έχουμε πολλούς ε, τομείς ε, που χρησιμοποιούν ε, στο έπακρο επαγγελματικό απόρριτο, για παράδειγμα συμβολιογράφοι, δικηγόροι. Ε, είναι διαφορετικοί επίση οι κανόνε που επικρατούν στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε και άλλου τομεί όπως είναι τα καζίνο, οι λογιστέ. Και εδώ χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω ανάλυση, αν θα θέλαμε κάτι να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να τα πετύχουμε τα πράγματα όπως τα επιθυμούμε. Να έχουμε μία αρχή δηλαδή η οποία θα επιτελεί το έργο της. Θέλουμε ασφαλώς να το εξετάσουμε αυτό. Δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις όμως. Δεν υπάρχει μία γρήγορη λύση η οποία θα μας ε, οδηγήσει ε, πάραυσα στην επιθυμητή κατάσταση. Θέλουμε λίγο χρόνο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Νίλς Φογκουσάν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της έκθεσης της Εποπτικής Αρχής των Τραπεζών του Απριλίου αυτού του έτους. Η Δανέζικη Τράπεζα υπήρχε είχε εμπλακεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για πολύ μεγάλα ποσά. Είναι μάλιστα ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της ιστορίας και πρέπει να σας πω ε, ξεπλάγει που η Εποπτική Αρχή είπε ότι ε, δεν υπήρχε παραβίαση δικαίου. Μιλάμε για 100 δις ε, ευρώ που ξεπλήθηκαν ε, από το 7, 2007 μέχρι το 2015. Οι δανέζικες αρχές προειδοποιήθηκαν πολλές φορές, δεν έκαναν τίποτα και έστειλαν ένα mail απλά στις άλλες τράπεζες αν όλα πάνε καλά, τους είπαν μια χαρά και δεν έγινε μετά τίποτα. Αυτό ήταν τεράστιο σκάνδαλο, όχι μόνο στην Δανία, αλλά γενικότερα στην ιστορία του ξεπλήματος. Η εποπτική αρχή είπε ότι δεν υπάρχει παραβίαση ενωσιακού δικαίου και αυτό κατά την άποψή μου είναι σκάνδαλο. Αν εδώ ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τότε δεν έχει και νόημα να υπάρχουν αρμόδιες αρχές ε, που ερευνούν την υπόθεση. Βεβαίως ε, αυτά όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο την ε, φήμη της, ε, της Οπτικής Αρχής Τραπεζών στη Δανία. Το θέμα είναι ότι πώς μπορούμε να έχουμε κανόνες οι οποίοι θα επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ε, παραδείγματος χάρη υπάρχει σαφώς σύγκρουση συμφερόντων όταν οι δανέζικες αρχές είναι εκείνες οι οποίες εγκρίνουν ή απορρίπτουν μια έκθεση ε, που λέει ότι δεν υπάρχει ε, παραβίαση ενωσιακού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ακριβώς προτίθεστε να αντιμετωπίσει το θέμα θα προτείνετε νέους, νέους κανόνες, διότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή ε, ε, εποπτική αρχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η εποπτική αρχή τραπεζών έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αυτό που ρωτάτε είναι τι κάναμε στο πλαίσιο της αναθεώρησης ε, στη νέα νομοθεσία. Ε, κατά κάποιο τρόπο έχουμε ενισχύσει τους ε, κανόνες έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και περισσότερες ρήτρες ασφαλείας για να μπορούμε να διασφαλίσουμε και την αντικειμενικότητα αποφάσεων που λαμβάνονται. Εγώ ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποια βήματα ε, για να ε, δούμε κατά πόσον όλα αυτά αρκούν ή κατά πόσον θα πρέπει να ξανασκεπτούμε κυβερνητικές δομές και τη δομή γενικότερα και της εποπτικής αρχής τραπεζών. Το ενωσιακό δίκαιο το ελέγχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μεταξύ άλλων και ίσως πρέπει να ε, υπογραμμίσουμε ότι η ε, εποπτική αρχή τραπεζών ε, μεταξύ άλλων θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη όσον αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αλλά το θέμα αυτό σίγουρα θα το προσέξουμε, θα το παρακολουθήσουμε. Ο κύριος Φεν για τους πράσινους. ο ένα αστιάκι έκανε ότι τώρα που μου δώσει το χρόνο να ήρθε και να μου μιλήσει και ο κύριος ε, Ότμαρ Κάρας, αλλά τέλος πάντων θα μιλήσει τώρα ο κύριος Κάζα. Ε, να κάνω κάποιες ε, σύντομε παρατηρήσεις, λέει ο κύριο Κάμπα. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι στην περίπτωση αυτή της Δανέζικης Τράπεζας η ε, εποπτική αρχή ε, στράφει περισσότερο κατά των αρχών της Δανίας. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε χρήση καλύτερων εργαλείων. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τελικά αυτή η περίπτωση ε, είναι μια περίπτωση όπου αξιολογείται μια τρέχουσα περίπτωση και κατά πόσον υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή των ε, κανόνων. Βέβαια, ε, στην περίπτωση αυτή δεν υπήρχε η ίδια αποτελεσματικότητα για να εξεταστούν προηγούμενες περιπτώσεις, το πώς ακριβώς ε, εφαρμόστηκε η ε, νομοθεσία κατά το παρελθόν. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι το εργαλείο δεν είναι αποτελεσματικό. Ο Σβέν. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, εφαρμογή της υφιστάμενης οδηγίας. Πριν από δύο χρόνια τα κράτη-μέλη έπρεπε να έχουν εφαρμόσει την τέταρτη οδηγία. Και θέλω να μας πείτε λοιπόν, πότε ξεκινήσατε τα διαδικασίες επί παραβάση. Και θα ήθελα να ξέρω πότε θα ολοκληρώσετε τον έλεγχο πληρότητα για την υλοποίηση της τέταρτη οδηγίας και πότε θα ολοκληρώσετε και τον έλεγχο ορθότητα για την εφαρμογή της τέταρτη οδηγία. και πότε επιτέλους θα εξασφαλίσετε πλήρη εφαρμογή της τρίτης οδηγίας, πολύ παλιά οδηγία πια. Η γερμανική μονάδα χρηματονομικής ευθείας είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στο συνολικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και σύμφωνα με τις ε, πληροφορίες που μας δίνει η Γερμανία δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί και αποτελεί και κίνδυνο ασφάλειας. Γιατί οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται από τις τράπεζες και από τις άλλες οντότητε που υποχρεούνται να χορηγούν α, τέτοια στοιχεία δεν χορηγούνται με τον τρόπο που πρέπει προ την αστυνομία. Και αυτό συνεπάγεται μεγάλο κίνδυνο ασφάλειας. Πείτε μας λοιπόν επακριβώς πότε επιτέλους θα καταφέρετε να υλοποιήσετε 100% την ε, ήδη φυστάμενη οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κίγκολτα. Να σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Για την τέταρτη οδηγία. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία επί παραβάση κατά όλων των κρετών μελών και όταν τέθησε το ερώτημα του κατά πόσον η τέταρτη οδηγία έχει ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της και τον ελεγχό της. Παραπέμψαμε δύο υποθέσεις στο δικαστήριο. Το θετικό είναι ότι, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, σήμερα έχουμε ολοκληρώσει τον έλεγχο πληρότητας και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι παρόλο που πήρε χρόνο και χρειάστηκε να ξεκινήσουν διαδικασίες επί παραβάση, υπάρχει πλέον μία πλήρης εικόνα. Αυτό επί το οποίο εργαζόμαστε ακόμα είναι κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουν ε, τύχει σωστή αξιολόγηση. Αυτό είναι μια διαδικασία εν εξέλιξη ακόμα. Και είμαστε σε επαφή με πολλά κρατημέλη και τη Γερμανία αλλά και άλλους για να ολοκληρώσουμε την αξιολόγησή μας. Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει 100% αλλά θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε το σύντομο δυνατό. Και θα δούμε κατά πόσον θα κινήσουμε τις διαδικασία. Ναι, πότε θα ολοκληρώσετε όμως ε, τη διαδικασία ορθότητας. Έχουν περάσει δύο χρόνια πλέον. Πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίε. Ενδεχομένω αυτό να πρέπει να γίνει σε φάσεις είναι η απάντηση. Γιατί πρώτον, κατά πρώτον θα πρέπει να έχουμε στο, στην διάθεσή μας το σύνολο της νομοθεσίας για να δούμε τι στέκει και τι δεν στέκει. Αυτό θα γίνει βαθμία ενδεχομένω. Αλλά δεν μπορούμε να σας πούμε σήμερα θα είναι σε δυο τρει μήνες. Εξαρτάται από το πόσο περίπλοκες θα είναι οι υποθέσεις που αντιμετωπίσουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ε, έχουμε πολύ δυνατή ομάδα. Έχουμε, είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας για μας. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν την πρώτη διαδικασία ήμασταν αισιόδοξοι θα πατήσουμε γκάζι στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ και έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας, λέει ο Πρόεδρος, και μας είπαν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο κ. Γκούναρ Πέκ έχει το λόγο και θα δώσω το λόγο και για δύο catch the Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θέλω να κάνω μία ερώτηση απευθυνόμενος κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ένας ε, τομέας ε, που μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τον έλαβε υπόψη της στην καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Αναφέρομαι στους μη κυβερνητικού οργανισμούς, στο ΜΚΟ, στους ΜΚΟ. Πέρυσι ο Κένετ Γουέν, ο επίτροπος από τη Μάλτα, ε, ζήτησε η νομοθεσία για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομοθεσία αυτή να επεκταθεί και στη ε, ΜΚΟ. Επειδή υπάρχουν ε, σαφείς αποδείξεις ότι οι ΜΚΟ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτή η άποψη βρίσκει απήχηση, γι' αυτό λοιπόν σας ε, ερωτώ γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα στον αγώνα της ε, κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, γιατί της ε, αγνόησε, και εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση της Ουγκάντα το πρόβλημα αυτό το εντόπισε ήδη πριν από πολλά χρόνια και το 2017 ε, θέσπισε ένα νόμο, ε, ένα νόμο κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ε, θα απαντήσω γερμανικά. Κοιτάξτε, εξετάζουμε όλες τις περιπτώσεις όπου έχουμε ενδείξεις ε, ότι μπορεί να υπάρξουν παράνομες ε, δραστηριότητες, ε, που υπάρχουν πάρα πολλές. Πράγματι, όσον αφορά τις ΜΚΟ, πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν στο ότι οι, οργανισ... οι ΜΚΟ ε, προβαίνουν σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε εντοπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε ε, σε επαφή με τη Μάνιβαλ και με άλλους ε, και ένα θέμα που θα το δούμε πολύ προσεκτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. For the catch the eye, Mr. για καλούνιας, από τους πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Δύο λεπτά, ε, δύο λεπτά. Ναι, θέλω να μάθω για το ρόλο των ε, διαδικτυακών τραπεζών, όπως ονομάζονται, με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες από την ε, λίγη εμπειρία που έχω. Δεν έχουν πολλές απαιτήσει, είναι πολύ χαλαρές, άνετα. Οι τράπες έχουν την εποπτεία και από εκεί έχουν και τη φήμη τους. Οι διαδικτυακές όμως είναι καθαρά θέμα αγοράς. Οπότε θέλω να ξέρω τι ρόλο έχετε εσείς αυτό. Και έπειτα για την Επιτροπή τον ρόλο των ε, μητρών επιχειρήσεων. Μερικές φορές σε κάποιες χώρες μέλη έχουμε καλά αποτελέσματα στις χώρες μέλη. Αντίθετα, άλλες φορές υπάρχουν πολύ χαλαρές διαδικασίες για να δηλωθεί κανείς το ότι δηλώνει και λοιπά. Πράγμα που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος στο σύστημα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Πριν τις απαντήσεις θα δώσω το λόγο και στον κύριο Βυζλάρο και μετά η απάντηση μια και έξω. Ευχαριστώ. Άκουσα την Επιτροπή. Πραγματικά θα πρέπει να είναι δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί έκανε ένα καλό βήμα να βελτιώσει την νομοθεσία και τώρα πρέπει να περιμένουν, κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Δεν προχωράμε. Έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με έγκλημα, μιλάμε για την νομιμοποίηση παράνομου χρήματος, σαν να είναι κάτι καθαρά τεχνικό και μόνο, αλλά δεν είναι γιατί πρόκειται και για εμπορία ανθρώπων, λαθρεμπόριο, από το οποίο ζημιώνονται πολλοί. Πρόκειται και για τους ανθρώπους, για τη ζωή των ανθρώπων. Μη συζητάμε λοιπόν έτσι σαν να πρόκειται για ένα καθαρά τεχνικό θέμα. Όχι, πρόκειται για τη ζωή των πολιτών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε εδώ να έχει έναν σύμμαχο. Δεν θα πρέπει να μπαίνουμε στην αμυντική. Όχι, αντίθετα. Να δράσουμε, να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Τι ακούσαμε σήμερα. Ακούσαμε ότι υπάρχει μια αξιολόγηση τον Ιανουάριο του 2020 και μετά μια έκθεση το 2022. Μα δεν είναι χρήσιμο αυτό. Τα πράγματα προχωράνε γρήγορα. Για να μην πω και ότι οι εγκληματίες προσαρμόζονται ακόμα πιο γρήγορα στη, στο νέο περιβάλλον. Να είμαστε λοιπόν σύμμαχοι μεταξύ μας. Ωραία, κάποιες χώρες ε, μέλη μπορεί να μη θέλουν Ωραία, ας μείνουν απ' έξω, ας προχωρήσουν οι υπόλοιπε. Συγκεκριμένα τώρα για την Επιτροπή. Δεν θα ήταν λογικό από πλευρά του Κοινοβουλίου να ληφθεί κάποια πρωτοβουλία. Μήπως αυτό θα βοηθούσε για να προθεθούν κάποια από τα θέματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τις προπτικές για να υπάρχει μια ενιαία αρχή που θα αντικαταστήσει το σημερινό θεσμικό πλαίσιο. Και δεύτερον, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, έχετε μονάδα για πληροφορίες, έχετε εντολή για να μπορέσετε να συλλαγετε πληροφορίες. Απαντήσεις και καταληκτικά σχόλια. Πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ναι, θα είμαι σύντομη. Για το πρώτο, για το Μητρό Επιχειρήσεων και τις σχετικές δυσκολίες. Ό,τι έχουμε κάνει με την οδηγία, το κοιτάμε και θα αλλάξουν τα πράγματα για να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι σε αυτό. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, να ξέρετε ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Και όπως ρώτησε και ο κύριος Κίγκολτ, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσει και διεθνώς. Για τη δεύτερη ερώτηση, Όντω έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά μέχρι τώρα στην προηγούμενη θητεία. Αλλά όχι μην νομίζετε ότι μόνο αναλύουμε. Κάναμε και την πέμπτη οδηγία η οποία προχωράει. Χρειαζόμαστε μια καλή βάση για να κάνουμε τη δουλειά μας. Για τελείως δεν θα πετύχει η νομοθεσία. Είναι σημαντικό λοιπόν να προχωρήσουμε με την μελλοντική αρχιτεκτονική, με ανοιχτό πνεύμα. Μην αρχίζουμε με το έτσι πρέπει να το κάνουμε, όχι να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε και τι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θέλει να κάνει η Επιτροπή και βεβαίω η συνεργασία μαζί σας πολύ σημαντική. Ο κύριος Κάμπα για τις διαδικτυακές τράπεζες. Είναι τράπεζες που υποβάλλονται σε εποπτεία όπως όλες οι τράπεζες, αλλά σωστά λέτε ότι δεν υπάρχει δέος επιμέλεια. είναι μια διασυνοριακή πρόκληση. Όντως ο κόσμος ε, διαμαρτύρεται γιατί η πρακτική διαφέρει ε, ανάλογα με το σε ποια χώρα βρίσκεται ο πελάτης και οι απαιτήσει είναι διαφορετικές και η ιδέως επιμέλεια του πελάτη διαφέρει. Οπότε μπορούμε να βάλουμε κατευθυντήριες γραμμές για την ε, εποπτεία, αλλά θα πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές. κάτι δεσμευτικό σίγουρα θα βοηθούσε. Για τη δεύτερη ερώτηση. Για τις ε, μονάδες πληροφοριών δεν έχουμε τέτοιες εμείς για οικονομικές πληροφορίες. Έχουμε εντολή σε ενισχυμένη συνεργασία ε, για ενημέρωση δεδομένων και πληροφορίες. Ξέρετε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών ε, περνάει από πολλούς περιορισμούς. Απλώς βλέπουμε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για διασυνοριακή συνεργασία. Αν υπάρχει κάποια ύποπτη κίνηση σε κάποιο σημείο, να έχουμε ένα κοινό σύστημα. Ωραία, ολοκληρώθηκε η σε αυτή. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει 23 και 24 Σεπτεμβρίου.